Καλημέρα σε όλους. Προτείνω να αρχίσουμε, διότι ο κύριος Μούλτερ που είναι και το πρόσωπο κλειδί για το πρώτο σημείο πρέπει να αποχωρήσει στη συνέχεια. Είναι εισηγητής μας για αυτό το ζήτημα. Και εντάξει, ευελπιστώ ότι θα καταφτάσουν κάποια στιγμή και οι υπόλοιποι συζητούμε για τη θέσπιση του συστήματος εποπτείας των σύνορων. Ε, χθες το βράδυ ο τριμερής διάλογος έλαβε χώρα από ό,τι ξέρω. Και θα ήθελα να σας ζητήσω κύριε Μούλτερ να πάρετε το λόγο πρώτος. Και στις 10 Ιουνίου θα ψηφίσουμε. Θέλουμε όμως να μας κάνετε ένα απολογισμό στο, για τον έκτο τριμερή διάλογο που έγινε. Κύριο Μόλντερ, ευχαριστώ Πρόεδρε χαίρομαι ε, που μου δίνετε το λόγο. Χθε ε, ελπίζουμε ότι ήταν ο τελευταίος ε, τριμερής διάλογος για το EuroSUR. Ε, σχετικά με την ενίσχυση της παρακολούθησης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν έχουμε ελεύθερη μετακίνηση των ατόμων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και ελπίζω ότι έχουμε πάρει, ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Ε, έγιναν διάφορες ε, διαπραγματεύσεις ε, επί τη βάση της αρχικής θέσης του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Αντίστοιχα έχουν γίνει παραχωρήσεις, έχει σημειωθεί πρόοδος. Το Κοινοβούλιο νομίζω μπορεί να δηλώσει ικανοποιημένο με αυτήν την συμφωνία. Το σημαντικό για εμάς είναι ότι θα πρέπει ε, να ε, κάνουμε κάτι για όσους πνίγονται στη Μεσόγειο προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη ε, η διάσωση αυτών των ανθρώπινων ζώων ε, είναι ε, προεξάρχον σημείο της δικής μας θέσης σε σχέση τώρα με τις διαπραγματεύσεις. Εμείς ισχυζόμαστε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με τρίτα μέρη. Χρειάστηκε όμως να υπαναχωρήσουμε ενώπιον του Συμβουλίου και, αν, ε, θα πρέ... Ε, και δεχτήκαμε για την σωστή λειτουργία του συστήματος ε, την ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων. Άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, τονίσαμε και πάλι τη σημασία της αρχής της μη επαναπροώθησης. Ε, ενσωματώθηκε αυτό μέσα στο κείμενο. Θα παραμείνει όμως αφιλεγόμενο το σημείο μέχρι το πέρας της διαδικασίας η συνθήκη πάντοτε μιλάει για παράτυπη μετανάστευση και παράνομους μετανάστες. Εμείς προτιμούμε τον όρο irregular, όχι παράνομο, παράτυπο, ε, παράτυποι μετανάστες και όχι παράνομοι μετανάστες. Αυτή ανέκαθεν ήταν η θέση μας. Ε, τροποποιήσαμε την φρασεολογία και μόνο στα τα άρθρα που συνάδουν με τη συνθήκη ε, διατηρήθηκαν. Ενισχύσαμε την δυνατότητα συνεργασίας ε, με ε, υφιστάμενα θεσμικά όργανα. Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Αλληλεία, για τη Θαλάσσια Ασφάλεια, τον Οργανισμό για την παρακολούθηση μέσω δορυφορικών εικόνων, παρακολούθησης επίσης της γης, δεν είναι διασυνδεδεμένα αυτά τα συστήματα με αυτό του Frontex. Εφ' θα είναι δυνατή η τακτική συνεργασία και συντονισμός όλων αυτών των υπηρεσιών. Το Κοινοβούλιο ε, πιστεύει ότι πρέπει να προαγάγουμε ε, τον ισχυρό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα παρακολουθήσει την υλοποίηση της συμφωνίας. Πρέπει επίση να ενημερώνεται η Επιτροπή και να εγκρίνεται κάθε πρόταση και τα κράτη-μέλη καταθέτουν τις προτάσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφαίνεται. Ε, αυτό είναι χαρακτηριστικό τη θέση του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά θα είναι συνάρτηση ε, των εξελίξεων της 6 ης Ιουνίου με την ε, ψηφοφορία. προς το παρόν συστήνω να προσπογράψετε και εσεί τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου. Πρόεδρος, προεδρεύουσα μάλλον. Ε, σας ευχαριστούμε για αυτήν την ε, συμφωνία. Ναι, ναι, ε, σωστά αυτά που λέτε και στη συνεδρία των συντονιστών ε, συμφωνήσαμε εχθές να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την έκφραση που αποφασίσατε και εσείς στον τριμερή, να μην μιλάμε για παράνομους μετανάστες, illegal migrants, παράνομη μετανάστευση είναι ένα όρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γιατί προβλέπεται και στη συνθήκη, όπω είπατε. Όταν μιλάμε όμω για μετανάστε, θα του χαρακτηρίζουμε παράτυπου και όχι παράνομου είναι ανα... Αναφέρονται πάρα πολύ συχνά αυτοί οι όροι και θέλουμε να αποφύγουμε αυτόν τον όρο, η regular. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν για την προετοιμασία της συμφωνίας. Είχα την εντύπωση όμως στη συνεδρία των συντονιστών εχθές πως ε, είναι κοινή θέση όλων, μπορούμε να δεχτούμε δηλαδή για το, τις μελλοντικές μας διαπραγματεύσεις ε, να υιοθετηθεί αυτός ο όρος. Υπάρχουν σχόλια παρακαλώ ο κύριος Μπρόνς, ε, παρακαλώ κύριε Μπρόνς. Ναι, ε, έφτασα στο τέλος. Δυστυχώς ακούσαμε για το τραγικό ε, ατύχημα σε όλα αυτά τα στις και τις Βάρκες ε, στη Μεσόγειο και τους θανάτους. Είναι λυπηρό όμως. Έχουμε και την αρχή της μη επαναπροώθησης. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η αρχή της μη επαναπροώθησης συμβάλλει στην απώλεια ζών διότι τι, θα περάσουμε το μήνυμα πως ε, αν έρχονται από μη ασφαλείς χώρες ε, σε καμία περίπτωση δεν θα επαναπροωθηθούν. Αν τους περάσουμε αυτό το μήνυμα ουσιαστικά τι τους λέτε. Λοιπόν, εάν εσείς προτίθεστε να αναλάβετε και να διατρέξετε αυτό το κίνδυνο θα ε, το πετύχετε και θα παραμείνετε στην Ένωση. Για την φρασιολογία δεν θα μου πούνε οι άλλοι ποιες λέξεις μπορώ να χρησιμοποιώ και ποιες όχι. Αυτοί που θα ήθελαν να περιορίσουν τους όρους ε, ουσιαστικά είναι οι ίδιοι που θέλουν να περιορίζουν και τη σκέψη μας. Ε, σας ευχαριστούμε κύριε Μπρόντ. Υπάρχουν άλλα σχόλια παρακαλώ. Ωραία. Θα γίνει η ψηφοφορία λοιπόν στις 10 ε, Ιουνίου. Ε, και προτού περάσουμε στο επόμενο σημείο θα ήθελα να σας ενημερώσω εξ ονόματος της κυρίας Αντωνέσκου που είναι η συγγήτρια για την οδηγία για την πρόσβαση σε ε, νομική αρρωγή, σε ποινικέ διαδικασίες. Στις 10 Μαΐου καταλήξαμε συμφωνία με το Συμβούλιο και έχουμε τώρα δύο φακέλους που ολοκληρώθηκαν και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 19 Ιουνίου στη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας. Λοιπόν... Ε, so... Λοιπόν... Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Φρανσουά Κχαϊπό, που είναι ο επόμενος ε, μιλητής μας ε, για την ε, διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολείται με τον αντίκτυπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών πιο συγκεκριμένα. Θα ακούσουμε την παρουσίαση έκθεση από τον κύριο Φρανσουά που είναι και ο ειδικός συγκητής του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών ε, μακροχρόνια μελέτη ε, επί του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού, από τα μέλη της Επιτροπής ε, και εκπροσώπους άλλων θεσμικών οργάνων για, το, για την Ιταλία, η Τουρκία και η Ελλάδα. Συμμετείχαν επίσης σε μια κοινή ομάδα εργασίας που μετήχε στην εκπόνηση αυτής της μελέτης και στις 27 Μαΐου δημοσιεύθηκε αυτή η μελέτη. Θα ήθελα λοιπόν Λοιπόν, να μας την παρουσιάσετε. Παρακαλώ θα σας δώσουμε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους ε, που με καλωσορίσατε εδώ. Θα ήθελα να σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση της θεματικής έκθεσης του 2013 που παρουσίασα ενώπιον του Συμβουλίου της, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΕ τη Δευτέρα και που εστιάζεται στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αποτέλεσμά της επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Ε, όπως αναφέρθηκε από σας, ε, ένα ολόκληρο χρόνο επεξεργαζόμουν αυτή την έκθεση. Ήρθα δύο φορές ε, στις Βρυξέλλες. Συναντήθηκα με βουλευτές, ε, με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Σε τέσσερις χώρες επισκέφτηκα επίσης για να κάνουμε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων ε, και την έρευνα που χρειαζόταν στην Τινησία και την Τουρκία. Ήταν η πρώτη μου επίσκεψη, δύο ε, γειτονικές χώρες όπου ε, ο αντίκτυπος των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την φύλαξη των συνόρων γίνεται αισθητό και σε επισκέφθηκα και την Ιταλία και την Ελλάδα από την άλλη πλευρά έχουν πολύ ευαίσθητα θα τα χαρακτήριζα σύνορα αυτές οι δύο χώρες και πρέπει να τα φυλάσουν. Ε, την περασμένη Δευτέρα παρουσίασα την μελέτη αυτή και πρόκειται για μια θεματική μελέτη, όπως σας είπα, που συνοδεύεται από ένα παράρτημα ε, όπου διεξοδικά παρουσιάζεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεσμικά όργανα ε, που υλοποιούν αυτή την πολιτική και έχουμε και τέσσερις εκθέσεις των χωρών στο παράρτημα επίση. Ικανοποιήθηκα όλο ιδιαίτερω από την απόκριση και τη συνεργασία που μου προσέφεραν οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, στις 21 Μαΐου έλαβα μία γραπτή ε, αντίδραση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το περιεχόμενο της μελέτης. Δεν συμφωνήσαμε σε όλα. Αυτό βεβαίως είναι φυσιολογικό για ένα διάλογο. Πάντως λαμβάνω σοβαρά υπόψη την έκθεση και χάρηκα πάρα πολύ για την αντίδραση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσα σε αυτή την έκθεση σημείωσα ότι πρόσφατη, πρόσφατα σημειώθηκε, ε, σημειώθηκαν εξελίξεις ε, στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνθηκε η συνολικότερη προσέγγιση για τη μεταναστευτική πολιτική κυρίως σε σχέση με την νομότυπη ε, μεταναστευσή. Επίσης, ως προς τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων έχει σημειωθεί πρόοδος ε, και κυρίως σε σχέση με τον Frontex και την αναθεώρηση του κανονισμού Frontex 2011 με το διορισμό ενός αξιωματούχου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Frontex καθώς και τη συγκρότηση του συμβουλευτικού φόρουμ του Frontex. Με τις αυξανόμενες αρμοδιότητες Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη μετανάστευση ε, δεν ε, είδαμε αντίστοιχε εγγυήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα πάντοτε. Όσοι πέφτουν ε, θύματα αυτή τη μεταναστευτική πολιτική και μιλάω για του ίδιου του μετανάστε. δεν είχαν αυτέ τι εγγυήσει, Κυρίω οι παράτυποι μετανάστε. παρότι ήταν σημαντικέ οι εξελίξει, λυπάμαι αλλά θα πρέπει να πω ότι στο πλαίσιο τη μεταναστευτική πολιτική, η παράνομη μετανάστευση θεωρείται θεωρείται, εξακολουθεί να θεωρείται ως μια ανησυχία για την ασφάλεια και αυτό καθοδηγεί την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και όχι την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης όπως εμείς θα επιθυμούσαμε. Μιλώντας για τη φρασιολογία που χρησιμοποιείται, αυτό είναι ένα ζήτημα ε, το οποίο σίγουρα θα πρέπει να το προβάλλουμε σε κάθε βήμα του διαλόγου για την ε, μετανάστευση και η χρήση όρων όπως ε, καταπολέμηση της παράνομης ή παράτυπης μετανάστευσης ε, θυμίζουν καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών. Ενώ όταν μιλάμε για παράτυπη μετανάστευση θα μπορούσαμε να καλύψουμε ένα ευρύτερο πεδίο των πολιτικών. Ε, αυτό επίσης ε, σχετίζεται με την ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος, να αντιλαμβανόμαστε ως ανθρώπους τους μετανάστες και άρα να αναγνωρίζουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Το Συμβούλιο ξέρω ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τέτοιε εκφράσεις σε παράνομη μετανάστες, σε παράνομη μετανάστευση στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, προτιμούμε, όπως ακούσατε και νωρίτερα, του όρου ε, παράτυπη μετανάστευση, παράτυπη μετανάστευση. Σε σχέση τώρα με τη μετανάστευση και την φύλαξη των εξωτερικών ε, συνόρων. Όλο ένα και περισσότερο η διάσταση τη ασφάλεια επικρατεί ε, και αντί να εστιάζουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα, επικεντρωνόμαστε, επικεντρώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προστασία των συνόρων από πλευρά ασφαλεία και όχι στην προστασία των δικαιωμάτων. Η εστιάζουμε λοιπόν στη μέσο επενδύσεων του Frontex για νέες ε, τεχνολογίες παρακολούθησης όπως το Eurosur που αναφέρατε ε, και εσείς ε, και το πρόγραμμα της Στοχόλμης που προβλέπει συντονισμό του Frontex για τις, για τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης δηλαδή για την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων αλλά προς το παρόν δεν συμβαίνει αυτό τουλάχιστον εγώ δεν το είδα. Στην Ελλάδα παραδείγματος χαρή όπου ελέγχονται οι μετανάστες στα σύνορα από την Ελλάδα για να ταυτοποιηθούν ως προς την υπηκότητά τους και να διευκολυνθεί ε, η ε, απομάκρυνσή τους. Αυτό ε, δεν συνέβη στα σύνορα, δεν εντοπίζονται οι ανθρωπιστικές ανάγκες δηλαδή. Το ίδια κατάσταση στην Ιταλία με τα κέντρα κράτησης που δημιουργήθηκαν για τους Τινήσιους και τους Αιγύπτιους στα πλαίσια και πρόσφατων ημερών διαπραγματεύσεων. Αυτά τα κέντρα σύντομης κράτησης ε, δέχτηκαν επίσκεψη από τον Frontex για τη συλλογή των ε, δεδομένων, όμως το κλιμάκιο του, ε, της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ και του Ερυθρού Σταυρού, του Ιταλικού, δεν έγιναν δεκτά στα αυτά τα κέντρα κράτηση και πρέπει να επιτύχουμε μια καλύτερη ισορροπία. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η κράτηση για να προετοιμαστεί η διαδικασία απέλασης θα πρέπει να είναι μέτρο ε, η έσχατη λύση. Ε, στα πλαίσια της έρευνας που έκανα ε, και βάσει της δράσης του Frontex βλέπω ότι για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων η συστηματική κράτηση των παρανόμων μεταναστών θεωρείται ως ένα θεμητό εργαλείο στα πλαίσια της διαχείρισης μεταναστευτικής πολιτικής από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ήταν η επιχείρηση στην Ελλάδα ο Ζεύς, ε, όπου ε, κρατούνταν αυτοί οι ε, παράνομοι μετανάστες, ενώ δεν ήταν απολύτως απαραίτητο. Θα ήθελα να σας παραπέμψω στην έκθεσή μου προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, του 2012, η περσινή μου έκθεση, δηλαδή γιατί το θέμα ήταν η κράτηση ακριβώς των παρανόμων μεταναστών. Εκεί τονίζω πως ε, η κράτησή τους ε, ποτέ ε, δεν έχει αποδείξει τον αποτρεπτικό σκοπό της για σκοπούς παράνομης μετανάστευσης. Για να μην παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κράτηση θα πρέπει να διέπεται από μια σειρά από κριτήρια, θα πρέπει να προβλέπεται από το δίκαιο, το διεθνικό δίκαιο, θα πρέπει να είναι απαραίτητη, λογική, αναλογική ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους. αν δεν πληρούνται αυτά τα κριτήρια, τότε η κράτηση παραβιάζει ε, το Διεθνές Δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της ε, διεξαγωγής μελέτης, είδα πολύ λίγες βιώσιμε λύσει να διερευνούνται είτε από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θεσμικό επίπεδο, είτε μεμονωμένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στι χώρες όπου μετέβην, είδα ότι είναι ανεπαρκή οι όροι κράτηση. Παραδείγματο χάρη δεν τηρούνται οικονομικές ή ουσιαστικέ νομικές εγγυήσεις για την κράτηση αυτών των ανθρώπων ε, που δεν έχουν καμία προοπτική απομάκρυνσης. Παραδείγματο χάρη όταν υποτιθέμενη χώρα προέλευση δεν του αναγνωρίζει, τότε παρατείνεται συχνά η κράτηση, ενώ δεν υπάρχει όμως ε, προοπτική απέλαση ε, και ω εκ τούτου η κράτηση δεν εξυπηρετεί κανένα στόχο στην ουσία πλέον και επίση η κράτηση των παιδιών. Η κράτηση των παιδιών ε, δυστυχώς απαντάται ε, σε πολλά σημεία σε αυτές τις τέσσερις χώρες ε, που επισκέφθηκα. Οι διαδικασίες επιστροφής επίσης, κυρίως των διευκολύνονται μέσω συμφωνιών επανεισδοχής, απέτυχαν ε, να παράσχουν τα απαιτούμενα ηχεία. Κατά τη διάρκεια της μελέτης παρατήρησε επίσης ότι είναι αυξανόμενη η εξίσταση. Ο έλεγχος δεν γίνεται στα φυσικά, στα πραγματικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βλέπουμε μια εξωτερική ανάθεση της εποπτείας των εξωτερικών ε, συνόρων και άρα μετακυλίεται η ευθύνη αποτροπή ε, της ε, παράνομης μετανάστευσης προς χώρες διέλευσης ή χώρες προέλευσης, κυρίως γειτονικές χώρες, μέσω της ανάπτυξης ενδογενών ικανοτήτων σε τρίτες χώρες με τρόπο ώστε να σταματήσουν να αναχαιτιστούν αυτά τα μεταναστευτικά κύματα. Παραδείγματο χάρη η συνεργασία ανάμεσα στο Frontex και την Τουρκία το 2012. Βεβαίω, η ανάπτυξη ενδογενών ικανοτήτων για ενισχυθούν οι υπηρεσίε φύλαξη των συνόρων και κατάλληλη κατάρτιση που εστιάζεται γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι αυτό βρίσκεται στον πυρήνα τη διαχείριση μεταναστευτική πολιτική, μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μεταναστών. Ε, δεν είναι κατά αυτό τη ε, τεχνολογική και τεχνική ε, συνεργασία για τον έλεγχο των συνόρων. Είναι ανησυχητική αυτή η εξωτερική ανάθεση προ άλλε χώρε και αυτό δεν συνοδεύεται από τα πρόσφορα εγγύα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, π.χ. τεχνική αρρωγή σε σχέση με το πώς ε, να παρασχεθεί πρόσβαση στη δικαιοσύνη ή στα αρμόδια εθνικά όργανα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για του μετανάστες ή για να έχουν αυτά τα όργανα την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τα απαιτούμενα μέσα προσωπικό με τρόπο ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ε, ε, κάνουν επισκέψεις στα κέντρα κράτησης ε, ώστε οι μετανάστες που χρειάζονται προστασία να εντοπιστούν και στη συνέχεια να έχουν την κατάλληλη μεταχείριση. Άλλη απόρρια του συστήματος διαχείρισης μεταναστευτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι οι χώρες που βρίσκονται γεωγραφικώς πώς στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σέγγεν όχι μόνο αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη φύλαξη των δικών του εθνικών συνόρων αλλά εποπτεύουν και φυλάτουν και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνήθω τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα είναι, ε, καλύπτουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις ε, και ε, για τα, αυτά τα συνοριακά κράτη αυτό συνιστά πάρα πολύ μεγάλο άχθος και ο Frontex πρέπει να τους επικουρήσει για την φύλαξη των σύνορων όμως παρατήρησα ότι είναι δυσανάλογα μεγάλο το αποτέλεσμα σε αυτά τα συνοριακά κράτη σε σχέση με τα, τις μεταναστευτικές δροές που φτάνουν στα σύνορά τους, κυρίως στην περίπτωση της Ελλάδας και ε, ε, επιμένω ότι κάποιοι παράγοντες όπως παραδείγματο χάρη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται εποχιακοί εργαζόμενοι και εργατικό δυναμικό που εύκολα μπορεί να πέσει θύμα εκμετάλλευσης, χαμηλής ειδίκευση στον τομέα της γεωργίας, εστίασης στον κατασκευαστικό τομέα. Εκεί η ανάγκη για εργατικό δυναμικό είναι υψηλή, όμως δεν αναγνωρίζεται τα, ε, ε, οι εργασιακές ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Αν έχουμε καλύτερους διάβλους μεταναστευτικούς, ακόμη και για θέσεις χαμηλής ε, ειδίκευσης, θα ανταποκρινόμαστε καλύτερες ανάγκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε μικρότερο αριθμό μεταναστών που παράνομα προσπαθούν να διέλθουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λιγότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Ο στόχος της σύντομη παρουσίασης μου είναι και να προβάλλω τα πορίσματα της αλλά και να αναφέρω ότι μέσα στην έκθεσή μου άμεσα απευθύνουμε ε, συστάσει σε θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και ελπίζω ότι αυτέ οι στοχευμένε συστάσει ε, ε, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας πιο ενός πιο συνεκτικού πλαισίου για την διαχείριση τη μεταναστευτική πολιτική και τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Σα ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει και παρατηρήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεσή σα. Ήταν μια πολύ σαφής ε, ενημέρωση για όλους μας. Έχουμε χρόνο για σχόλια και ερωτήσεις. Η κυρία Ρομέρο Λόπες, Κάρμεν, έχεις το λόγο, είσαι η πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ε, και ίσως θα ήταν καλύτερο να είχατε εμβαθύνει λίγο περισσότερο στην ε, κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα κέντρα κράτησης στις ε, χώρες που βρίσκονται σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, όπως είπατε, υπάρχουν προβλήματα προβλήματα δικονομικών εγγύσεων. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στα σύνορα των ε, χωρών της Νοτιού Ευρώπης έχουμε μικρά γκουαντάναμο γιατί είναι απαράδεκτο να υπάρχουν παράτυποι μετανάστες ή αιτούντες ε, άσυλο γιατί όλοι είναι αναμειγμένοι και να διαμένουν σε κέντρα κράτησης και να περνούν εκεί τρεις ως έξι μήνες χωρίς να έχουν απολύτως καμία δυνατότητα πρόσβαση σε κανένα απολύτως δικαίωμα δικαιώματα ε, τα οποία παλαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και πολύ συχνά σε πολλές ε, χώρες μετά από τους έξι μήνες τους αφήνουν ελεύθερους και τελικά επιστρέφουν, κρατούνται και πάλι για άλλους έξι μήνες. Αυτή η κατάσταση είναι απολύτως ε, παράδεκτη. Δεν είναι φυσιολογική κατά κανέναν τρόπο. Δεν είναι μια κατάσταση που θα πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να θεωρούν ότι είναι συμβατή με τις αξίες και τα δικαιώματα που ασπίζουμε. Είναι εντελώς απαράδεκτο. Αυτά τα κέντρα κράτησης, εμείς είδαμε τι γίνεται στην Ελλάδα για παράδειγμα ή τι γίνεται στη Μάλτα. Στην Ελλάδα, στη Μάλτα και στην Ισπανία. Ε, δεν είναι δυνατόν η κατάσταση αυτή να παραταθεί περαιτέρω. Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί σε πολλέ χώρε δεν έχουν απολύτω καμία πρόσβαση σε αυτά τα κέντρα κράτηση. Ε, δεν υπάρχουν καθόλου, δεν έχουν δυνατότητα νομικής υπεράσπιση. Δεν έχουν ε, δικηγόρους. Άρα υπάρχουν τεράστια νομικά κενά εδώ δεν βρισκόμαστε σε περιπτώσεις ε, πολέμου. Είμαστε χώρες υποδοχής ή όπως η Συμφωνία του Δοβλίνου. Αυτές οι χώρες είναι υποχρεωμένες να υποδεχθούν αυτούς τους ανθρώπους. Άρα δεν είναι μόνο το νομικό κενό, αλλά οι χώρες αυτές με τις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν τα τεράστια ελλείμματα και τα χρέη δεν μπορούν να υπομισθούν αυτή την κατάσταση. Χαίρομαι που οι τα Ηνωμένα Έθνη δείχνουν ένα ενδιαφέρον για αυτό το φαινόμενο της ε, παράνομης μετανάστευσης, αλλά θα πρέπει να βρεθεί μία λύση. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη σε αυτά τα κέντρα κράτησης και θα ήθελα πραγματικά να δείξετε ενδιαφέρον, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ε, μη κυβερνητικών οργανισμών σε αυτά τα κέντρα κράτηση, ούτω ώστε αυτοί οι πολίτε να έχουν τα ίσα δικαιώματα με του υπόλοιπου Ευρωπαίου πολίτε. Ο κύριο Παπα-Νικολάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρεπό για την ε, εισαγωγή του, για την παρουσίασή του και επιτρέψατε μου να κάνω αυτή την παρέμβαση στα ελληνικά και αυτό για πολλούς λόγους. Παρακολούθησα με πολύ προσοχή τα όσα αναφέρατε και μελέτησα το κείμενό σας με πολύ προσοχή. Και σέβομαι απολύτως το ρόλο σας και το γεγονός ότι η έκθεσή σας στοχεύει στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υπηκών των τρίτων χωρών και σε αυτή τη βάση βεβαίως με πολύ ε, προσοχή ε, διαβάζουμε τις παρατηρήσεις όπως αυτό το πράττουμε και για την έκθεση και στην αντίστοιχη έκθεση που έχει κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Fundamental Rights Agency, ε, και ε, σε κάθε ευκαιρία, με κάθε ε, αφορμή και με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που υπάρχουν, τις οποίες αναφέρετε όπως είδα και εσείς, και πολλές αποστολές που έχουν γίνει, και να διευκρινίσω ότι αντίστοιχε αποστολέ κάνει και αυτή η Επιτροπή. Και αυτή η Επιτροπή ε, είχε τη δυνατότητα να δει τι συμβαίνει και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Ελλάδα και θα πάμε και στην Ισπανία τώρα για να δούμε ε, τι συμβαίνει με τις επεμβάσεις της Frontex εκεί στα θαλάσσια, στη θάλασσα. Δεν άκουσα καθόλου στην εισαγωγή σας να αναφέρεστε στο smuggling από τις αποστολές που και εμείς έχουμε κάνει και έχω την αίσθηση ότι είναι κοινό τόπος αυτός ένας τεράστιος αριθμός η συντριπτική πλειοψηφία των υπηκών των τρίτων χωρών που φτάνουν στην Ελλάδα και την Ιταλία αναφέρομαι σε αυτές τις χώρες ιδιαιτέρως γιατί αυτές αναφέρεται και στην έκθεσή σας έρχονται με τη βοήθεια διακινητών και δεν, επειδή ο ρόλος ο δικός σας είναι ακριβώς αυτός, να βλέπετε συνολικά τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν είδα να δίνετε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι την περίοδο, την κρίσιμη με τις αναταραχές στη Βόρεια Αφρική ε, από, τον, από την Αφρική και να φτάσουν στη Λαμπεντούζα είχαν συγκεκριμένες οδηγίες πολλές φορές από τους διακινητές να Να βουλιάζουν τα πλοιάρια για να, τρέχουν, για να σπέβδουν οι αρχές της Ιταλίας αλλά και της Ευρώπης να κάνουν ε, επέμβαση και να τους διασώσουν με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο και με βάση τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους αυτούς. Το δεύτερο το οποίο δεν άκουσα στην αναφορά σας είναι ότι ειδικά για τις χώρες που αναφέρετε, που επιτρέψτε μου να πω Νιώθω ενοχλημένος όταν για την Ελλάδα, για παράδειγμα, γράφεται ότι πήγα σε ένα κέντρο, είδα ότι χωρούσε 28, είναι 26, αλλά κάποιο μου είπε ότι δεν ήταν τόσοι και ήταν παραπάνω. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ fact-finding mission. Και κάπου εκεί αισθάνομαι ότι ε, ενδεχομένως υπάρχει ένα στοιχείο υπερβολής. Το ίδιο για την Ιταλία. Διαβάζω τι παρατηρήσει σα. Οφείλω να σας πω ότι η Επιτροπή μας βρέθηκε στην Ιταλία αμέσως μετά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης. Βρεθήκαμε εκεί ε, τον, το, το, το χειμώνα, τον, τον τέλος Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, του 2011 και στην, ε, στην αποστολή αυτή είδαμε και πολλές βελτιώσεις στην προσπάθεια των χωρών αυτών, Τι, των, των κέντρων και των, των θέσεων υποδοχής των υπηκών τρίτων χωρών. Είδαμε την προσπάθεια των Ιταλικών αρχών να σεβαστούν τα δικαιώματα των, ε, ανθρώπων που έφταναν στην, ε, στην χώρα τους, όπως βεβαίως και την προσπάθεια των αρχών να μεταδώσουν στους Ιταλούς πολίτες, στους Ευρωπαίους πολίτες και το αίσθημα της ασφάλειας ότι αυτός ο τεράστιος όγκος αφήξεων δεν θα επηρεάσει την κοινωνική συνοχή της χώρας. Και αυτή η απειλή υπάρχει σε, και, και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Να αναφερθήκατε στο, στην ΕΑΖΟ. Η ΕΑΖΟ είναι μια καινούργια υπηρεσία, η οποία και αυτή προσπαθούμε να την υποστηρίξουμε και να, να αναπτυχθεί με ταχύτητα και να ενισχυθεί και σε ό,τι αφορά το έμψυχο δυναμικό της, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή τις μεγαλύτερες δυνατές ε, δυνατότητες για να, για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Ε, δεν, δεν βλέπω όμως και κάποιο σχολιασμό από την πλευρά σας ότι είναι σημαντικό ότι τη φτιάξαμε την ΕΑΖΟ. Είναι, τελειώνω κυρία Πρόεδρε. Είναι σημαντικό ότι μπορέσαμε και δημιουργούμε τις δομές και με το πακέτο ασύλου που τώρα ε, ψηφίζουμε και αποφασίζουμε την ανανέωση και την αναθεώρησή του ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικές βελτιώσεις κυρίως στο θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κλείνω κυρία Πρόεδρε. Ένα τελευταίο, ε, ένα τελευταίο νούμερο θα δώσω και με συγχωρείτε που κάνω κατάχρηση του χρόνου, αλλά είναι υποχρέωσή μου να το κάνω, γιατί αισθάνομαι ότι οι προσπάθειες που κάνουν οι χώρες αυτή τη στιγμή, που είναι ε, προσπάθειες που αφορούν όλη την Ευρώπη, ε, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη έκθεση και υπάρχει μια μονομέρεια σε κάποια, σε κάποια από τα σχόλια, τα οποία αδικούν τις χώρες αυτές. Ένα τελευταίο λοιπόν μέγεθος, γιατί στην έκθεσή σας, κύριε Κρεπό, δεν βλέπω πολλά νούμερα και θα ήθελα να δω περισσότερα. Το 2012 η Ελλάδα έκανε στην Τουρκία 292 αιτήματα για να γυρίσουν πίσω ομάδες υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είχαν νόμιμο έρισμα για να μείνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, που αφορά 20.464 μετανάστες και τελικά έφτασαν στην Τουρκία, για να μην σας κουράζω, μόνο 113. Πιστεύετε ότι όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή 20.300 είναι σε κέντρα κράτησης. Δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Όλοι αυτοί είναι στην, είναι, έχουν τη δυνατότητα, της, οι περισσότεροι από αυτούς κυκλοφορούν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και είναι καθήκον όλων μας να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε όσους μπορούν να είναι νόμιμοι και να αποκτήσουν έρισμα είτε με, ε, με αίτημα για διεθνή προστασία ή άσυλο είτε ότι, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να μείνουν. Οι υπόλοιποι όμως πρέπει και με τη συνεργασία των τρίτων χωρών να προωθηθούν προ τα εκεί. Και αυτό συμβαίνει και με το Πακιστάν που κάναμε συμφωνία και βεβαίως είναι υποχρέωση νομίζω για να σεβαστούμε τα δικαιώματα όλων αυτών των ανθρώπων, να συνεργαστούμε με τις τρίτες χώρες στα πλαίσια των συμβάσεων σε διμερές και διεθνές επίπεδο που καταρτίζουμε, οι οποίες αν μη τι άλλο προσπαθούμε να εφαρμόζονται και οι οποίε είναι μια προστιθέμενη αξία. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό δεν το θε... ενώ το αναφέρετε και λέτε ότι μπορεί να γίνει, μα λέτε ότι το πάμε, πάμε του ελέγχου και εκτό των συνόρων μα και ότι προσπαθούμε να, συνεργαστούμε με τι τρίτε χώρε, ω αν να έχουμε μια διάθεση να μην σεβαστούμε τόσο πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακριβώ το αντίθετο. Είναι ο μόνο τρόπο όμω για να το κάνουμε. Συγγνώμη, I'm sorry, Madam Chair, for, for, for taking more time, but this is Πάμε κυρία Πρόεδρε που πήρα περισσότερο χρόνο, αλλά είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Όντω είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινιστούν τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό για όλους μας. Γι' αυτό καλό είναι να ακούσουμε όσο το δυνατόν τα περισσότερα μέλη και να έχουμε και έναν διάλογο, δηλαδή να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από όλους οι ερωτήσεις να περιοριστούν στα δύο λεπτά, έστω και αν αυτό δεν είναι εύκολο, το γνωρίζω. Αλλά θέλω να μιλήσουν όσο το να περισσότερα μέλη μας. Κυρία Βίξτρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Κρεπό για την τόσο πλήρη ενημέρωσή του. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή φέρνει ελπίδα και έμπνευση ε, στην, ε, στην Επιτροπή μας. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ, αλλά να χρησιμοποιήσω όμως και τα υπόλοιπα 99 δευτερόλεπτα που έχω στη διάθεσή μου. Να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα έγκαιρη και επίκαιρη η, η ενημέρωση αυτή. Έχουμε ε, προχωρήσει στην νομοθεσία μας. Ασχολούμε, θα ασχοληθούμε τώρα με την παράνομη μετανάστευση. Ήμουνα ε, εισηγήτρια σε μία έκθεση για την ε, για τη μετανάστευση και για το πώς κάποια επαγγέλματα όπως οι οικιακές βοηθοί, ή βοηθήματα για τα παιδιά κτλ. θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό που είπατε, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διατύπωση ότι πρέπει να αλλάξει ο όρος παράνομος, διότι κανείς δεν είναι παράνομος, μπορεί να είναι, να είναι παράνομη βάση η νομοθεσία, ε, να παραβιάζει μάλλον την νομοθεσία για να είναι στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να πούμε ότι είναι παρατυπία ενδεχόμενα ή ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Άρα το θέμα δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρω... Ε, αφορά όλο τον κόσμο και ίσως ε, και τα Ηνωμένα Έθνη θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και πιστεύω ότι η παρέμβασή σας σήμερα χρήζει ε, σεβασμού και θα ήθελα να τονίσω και ελπίζω ότι και οι υπόλοιπε εκθέσεις που θα πούμε θα είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος. Κυρία Λάμπερτ, ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τα όσα ακούσαμε και είδα ότι αυτό το οποίο αποτελεί ένα κατευθυντήριο, μια κατευθυντήρια γραμμή, ένα, ένα, έναν ιστορία άδνης είναι ε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Ε, είπε η συνάδελφος για το πόσο επίκαιρη είναι η παρουσίαση αυτή, αν θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, και μιλήσαμε και για την εφαρμογή, αλλά κάποια από τα παραδείγματα τα οποία μας δώσατε, ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, η Frontex που έχει πρόσβαση ε, σε, κάποια, σε, κάποια, σε κάποιους θεσμούς, όχι όμως η υπατή αρμοστία. Αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί. Ε, ενώ υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διορθωθούν. Μήπως θα μπορούσατε να πείτε κάτι παραπάνω για, τα, για αυτά που είπατε για την παρακολούθηση των επιστροφών των απελάσεων. Να μας πείτε τι ακριβώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει εδώ. Τι θα Αυτό νομίζω θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μας είπατε ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν, δεν ξέρουμε τι εναλλακτικέ υπάρχουν όσον αφορά την κράτηση ε, περιμένοντας ε, να επιστρέψουν στη χώρα τους οι μετανάστες. Ποιες είναι αυτές είναι οι εναλλακτικέ λύσεις ε, που έχουν στη διάθεσή τους αυτοί οι μετανάστες. Στο Βέλγιο, παραδείγματο χάρη, κάποια άτομα τα οποία κρατούνται, συλλαμβάνονται, τους ε, αποστέλλεται μία επιστολή με την ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να αποχωρήσουν, να απομακρυνθούν από τη χώρα. Αυτή είναι η, η εναλλακτική λύση. Αν ναι, δεν είναι ουσιαστική λύση αυτή. Κύριε, κύριε Κρεπό, πρέπει... έχω την αίσθηση ότι δεν σας απασχολεί μια ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Είπατε ότι ένας έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα της κοινότητας δημιουργεί προβλήματα. Εγώ το αντίθετο πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι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 Ε, πρόσφατα μίλησα με συναδέλφους από τη Γερμανική Βουλή οι οποίοι έκαναν μια αποστολή στα στρατόπεδα αυτά κράτησης στην Ελλάδα και οι περιγραφές τους ήταν ε, πολύ πιο άσχημες όσον αφορά τη δεινή κατάσταση των ε, προσφύγων που γυρίζουν στο δρόμο των Αθηνών ή βρίσκονται σε αυτά τα κέντρα κράτησης. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να επιλέξω μια άλλη προσέγγιση. Πολύ συχνά λέμε ότι εκείνοι οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη μέσω διακινητών και ε, ποτέ δεν διατυπώνεται τόσο ρητά, αλλά πάντοτε αυτό υπονοείται, είτε είναι ενδυνάμοι εγκληματίες ή επιθυμούν να απολαύσουν τις ε, κοινωνικές παροχές σε αυτές τις χώρες και είναι ένας παράγων υψηλού κόστους στις χώρες μας. Ε, τι γίνεται όμως με τους πρόσφυγες οι οποίοι δεν καταλήγουν στην Ευρώπη αλλά πάνε στην, παραμένουν στην Αφρικανική Ήπειρο. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Και θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι όλοι όσοι πραγματικά επομίσονται όλους αυτούς τους κινδύνους, βρίσκονται υπό τεράστια πίεση γιατί δεν ε, πρέπει μόνο να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τη διαβίωση για τους ίδιους, αλλά πιέζονται από το γεγονός ότι θα πρέπει να βρουν χρήματα για τις οικογένειές τους για να χρηματοδοτήσουν τους διακινητές. Και αυτή είναι τεράστια οικονομική επιβάρυνση. Ε, ε, λέμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια δημογραφική μεταβολή και πολλούς τομείς δεν υπάρχει ειδικευμένο δυναμικό. Στη Γερμανία ε, γίνεται μια συζήτηση να έρθουν συναλλευτές από την Κίνα. Ε, και επίσης ε, υπάρχει στα νοικοκυριά μεγάλη ζήτηση για προσωπικό στις οικογένειες. Αλλά και αντί να εξετάσουμε λοιπόν σε ποιο βαθμό μπορούμε να δώσουμε μια προπτική σε αυτούς τους ανθρώπους στην Ευρώπη και αντί να το κάνουμε και να προσπαθήσουμε να τους αφομοιώσουμε, να ζητάμε από την Κίνα νοσηλευτικό προσωπικό, θεωρώ ότι αυτό είναι εντελώς ε, παράλογο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και μία νέα συζήτηση. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο θέμα της Ιταλίας. Ενδεχομένως υπάρχουν ορισμένα τέτοια ωραία και ε, προοδευτικά κέντρα κράτησης ε, στην Ιταλία. Αλλά εν μέρει άρχισε η Ιταλία να κλείνει αυτά τα κέντρα ε, και λέγεται ότι του πληρώνει στον κάθε πρόσφυγα 500 ευρώ για να φύγει από τη χώρα ή για να βρει μια άλλη λύση. Θεωρώ ότι συζητώντας για το θέμα των προσφύγων ε, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια πιο ουσιαστική λύση για αυτούς τους ανθρώπους εάν ε, μπορούσαμε να αλλάξουμε τη συνθήκη του Δουβλίνου αυτό θα ήταν πολύ θετικό γιατί ε, είναι συνέπεια αυτής της πολιτικής και έχει σαν αποτέλεσμα αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή στα κέντρα κράτησης στα σύνορα της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Κρεπό για την έκθεσή σας. Νομίζω ότι πραγματικά αποτελεί μια σύνοψη ε, και αναλύσεων ε, και παρατηρήσεων που ούτως ή άλλως και τα μέλη της Επιτροπής μας είχαν κάνει σε διάφορες αντιπροσωπείες, σε επισκέψεις όταν διαβάζαμε τα, τις εκθέσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το βασικό όμως ε, θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για την κατάσταση των συνόρων, ε, με βέβαια κάποια θέματα τα οποία είναι πιο σημαντικά για την κράτηση, παραδείγματο χάρη, ή για, τον, ε, για, την, για την ανάθεση κάποιων αρμοδιοτήτων και κάποιων υπηρεσιών σε κάποιους άλλους. Η έκθεση αυτή όμως παρουσιάζεται από ό,τι κατάλαβα σε όλα τα μέλη, σε όλα τα κράτη ε, ε, μιλάμε για τα Ηνωμένα Έθνη και ε, εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει πάντα τι πρέπει να γίνει, ποιο είναι το δίκαιο κτλ. Και εκεί ε, εκπονήθηκε η έκθεση αυτή και εκεί θα εξεταστεί και θα σχολιαστεί. Αυτό είναι το νέο στοιχείο και εγώ θέλω να ξέρω αυτή η έκθεση πώς θα ζήσει, πώς θα κυκλοφορήσει, ε, πώς θα ειδωθεί από, τις, από τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, τι συνέχεια θα δοθεί σε αυτή την έκθεση εμείς σαν βουλευτές θέλουμε να γίνουν σεβαστά να, τα δικαιώματα, το δίκαιο των ανθρώπων αυτών. Ε, εσείς τι θα κάνετε στα Ηνωμένα Έθνη έτσι ώστε να βελτιωθεί το κράτος δικαίου στα σύνορα της Ένωσης. Ευχαριστώ. Κυρία Γκυγιώμου, θα είμαι πολύ πιο σύντομη από ό,τι προβλέπετε, διότι δεν έχω να ε, να προσθέσω ή να αφαιρέσω ε, σε αυτά που είπε η κυρία Φλότρο. Όντως ε, και εγώ τα ίδια ήθελα να πω όσον αφορά τη συνέχεια που θα δοθεί σε αυτή την έκθεση και όσον αφορά τα κράτη-μέλη, διότι κάνετε κάποιες συστάσεις, αλλά και για το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια, η, ποιο, ποιο, ποια θα είναι η συνέχεια και ποιο είναι το βάρος αυτών των παρατηρήσεων παρατηρήσεις που ούτως ή άλλως επαναλαμβάνουν λίγο πολύ και αυτές που έχουμε κάνει και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. θα ακούσουμε και για τις συστάσεις αυτές. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ έχω ορισμένες ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την έκθεσή σας και λυπούμε που άργησα λίγο, αλλά μπόρεσα έτσι να το κοιτάξω. Και πράγματι, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, είναι μια πολύ καλή σύνοψη των όσων και εμείς παρατηρούμε στα εξωτερικά μας σύνορα. Και θα ήθελα να επενθυμίσω ότι βεβαίως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς συμμετέχουμε στην ε, θέσπιση των νόμων που διέπουν τα εξωτερικά σύνορα. Έχουμε συμφωνίες ε, υποδοχής, ε, συμμετέχουμε στη διαδικασία, στη, στη θέσπιση νόμων για τη χορήγηση ασύλου κλπ. Το ερώτημά μου αφορά την εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των συνόρων σε άλλες χώρες. Ε, βλέπετε εκεί καθόλου νομικά προβλήματα, γιατί προφανώς εκεί λειτουργούμε εκτός της δικής μας ε, επικράτειας. Επίσης, όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για τα κέντρα κράτησης, δεν ξέρω, διερωτώ με κατά πόσο ε, έχετε κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις για το θέμα της κράτησης και της σχετικής οδηγίας. Επίσης, όσον αφορά τα κονδύλια για το επόμενο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, τι θα γίνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ελέγχους των συνόρων. Τι θα πρέπει, πιστεύετε, να συμβεί άμεσα στα σύνορα, τους, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των μεταναστών. Και κάτι άλλο. Έγινε μια συζήτηση χθε για το Συμβούλιο, για την διάσωση ανθρώπινων ζώων στη θάλασσα, τι γίνεται με αυτό και ποιος είναι υπεύθυνο. Και οι χώρες μέλη λένε ότι είναι δική τους ευθύνη και δεν θα πρέπει να συμπεριφθεί αυτό στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά εσείς θεωρείτε ότι θα μπορούσε να διαδηματρήσει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίζοντας ένα δίκαιο για τη διάσωση ζώων στη θάλασσα. Επίσης για μέτρα για την επιστροφή. Πότε θα γίνει αυτή η έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την επιστροφή μέσω, των, μέσω της ε, Frontex. Ε, θα θέλω να μας ε, διευκρινίσετε την ημερομηνία, παρακαλώ. Ο κύριος Τενταφυλίδης είναι ο επόμενος ομιλητής. Ο Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω τον ομιλητή μας για την ε, πάρα πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίασή του. Ε, θέλω να απολογηθώ γιατί δεν έχω διαβάσει την έκθεσή του και επομένως δεν ξέρω εάν στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται και εισηγήσει για επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Νομίζω ότι πολλοί από εμά έχουμε την τάση να απλώς να περιγράφουμε τα προβλήματα, να περιγράφουμε την κατάσταση, αλλά δεν προτείνουμε λύσεις στα προβλήματα. Για παράδειγμα το ερώτημα του κυρίου για τους μετανάστες που δεν δέχτηκε η Τουρκία να επιστραφούν από την Ελλάδα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι προτείνουμε, τι εισηγούμαστε. Το ερώτημα του κυρίου Κλέης για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται εκείνοι οι μετανάστες κατά την περίοδο που αναμένουν μέχρι να επιστραφούν στις χώρες καταγωγής ή στις χώρες πρώτης εισόδου στην ε, Ευρώπη. Άρα εκείνο που θα ήθελα να δω και απολογούμε αν υπάρχει και δεν το είδα είναι προτάσεις για λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Ε, Mr. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπρόνς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο μιλητής ε, κατέκρινε την κράτηση παράνομων ή μάλλον παράτυπων μεταναστών. Ακούσαμε από τον επικεφαλής της Frontex πέρσι ότι οι παράνομοι μετανάστες κρατούνται μόνο προσωρινά και στη συνέχεια είτε τους επιτρέπεται να παραμείνουν μόνιμα στη χώρα, είτε τους αρνείται η παραμονή στη χώρα και τους ζητείται να αποχωρήσουν μέσω ενό εγγράφου. Βεβαίω δεν επακούν πάντοτε σε αυτή την οδηγία. Είπε ότι αν κάνουμε πιο εύκολη την νόμιμη μετανάστευση θα υπάρξουν λιγότεροι παράνομοι μετανάστευσης αλλά βεβαίω αν το επιτρέψετε οι άνθρωποι θα το κάνουν χωρίς ε, άδεια. Ε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να απορροφήσουμε όλους τους ε, μετανάστες. δεν μπορούμε, δεν είναι δυνατό να τους στεγάσουμε και τους παράσχουμε κατάλληλη τροφή. στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. ε, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να, δεν θέλουν να γίνουν κατ' ουσία Ευρωπαίοι. Εάν έρθουν περισσότεροι παράνομοι μετανάστες στην Ευρώπη, ε, το τον κίνδυνο να μετατρέψετε κομμάτια της Ευρώπης στον τρίτο κόσμο, όπως έγινε στο Λονδίνο πριν από μία εβδομάδα. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Παπανικολάου να πάρει το λόγο δεύτερη φορά γιατί είναι ο μόνος ο οποίος σχολιάζει από το ΕΛΚ και εφόσον είναι Έλληνας και η Ελλάδα αναφέρθηκε κατά επανάληψη θα δώσω το λόγο για λίγη ώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να διατυπώσω μια ξεκάθαρη ερώτηση. Μετά από όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν από τους συναδέλφους και λόγω του γεγονότος ότι έγινε ειδική μνήα για ορισμένες χώρες, ε, την Ελλάδα και την Ιταλία συγκεκριμένα, το ερώτημα είναι το εξής και θα ήθελα εδώ μια ξεκάθαρη απάντηση. Βλέπετε ως ε, συμπέρασμα της σημερινής ε, συζήτησης ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε έλλειψη, έλλειμμα αλληλεγγύης και σωστού επιμερισμού. Δηλαδή ή το σύστημα λειτουργεί καλά και είναι το απολύτως κατάλληλο και ενδεδειγμένο ή υπάρχει ανάγκη να επικριθούν ορισμένες χώρες μέλη γιατί δημιουργούν ακριβώς κενά σε, αυτό το, σε αυτή την ελεγγύη, αν θέλετε, και το σύστημα σωστού επιμερισμού των ευθυμονών. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τώρα έχετε περίπου 15 λεπτά να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις και να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ζωντανή συζήτηση. Ε, βλέπω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι ε, υπάρχει γνώση σε αυτή την αίθουσα ε, και εξειδίκευση θα τολμούσα να πω και ότι τα θέματα αυτά ζητούνται ε, κάθε μέρα εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται, δεν πρόκειται να απαντήσω σε κάθε ερώτηση με τη σειρά που ετέθη, θα δώσω μια συλλογική απάντηση. Αυτό το οποίο ζητάω σε αυτή την έκθεση είναι να γίνει μια μετατόπιση ε, ε, στον τρόπο με τον οποίο να γίνονται τα πράγματα. Δεν λέω ότι η Frontex πρέπει να υπάρχει ή ο έλεγχος στο εξωτερικά ε, των, των, των, των συνόρων της κοινότητας δεν πρέπει να γίνει. Απλώς λέω ότι υπάρχουν κάποιες αποστολές που έχουν δοθεί σε κάποιους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αποστολές αυτές είναι σωστές. Το πρόβλημα είναι πώς υλοποιούνται αυτές τις αποστολές, πώς εκτελούνται οι αποστολές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στις περισσότερες χώρες ε, οι μετανάστες ε, αποτελούν ε, ευαίσθητο μεν πληθυσμό, αλλά κάτω από στη σειρά ε, άλλων γυναίκες, ε, ομοφιλόφιλους ε, και όλοι αυτοί έδωσαν κάποιες μάχες, οι αυτόχθονες παραδείγματος χάρη και αυτό ισχύει για τους Βορειοαμερικανούς και τα λοιπά, τέλος πάντων έδωσαν μάχες και κέρδισαν τα, το σεβασμό των δικαιωμάτων τους, κινητοποιώντας τους πολιτικούς και κερδίζοντας σε δίκες. Όμως οι μετανάστες έχουν κάποια, είναι τα, φτάνουν στα δομικά όρια της δημοκρατίας, της δημοκρατίας μας, διότι οι μετανάστες δεν εκπροσωπούνται πολιτικά, στο πολιτική, στην πολιτική σκηνή, δεν μετράνε. Και δεν αναφέρω, δεν είναι θέμα των πολιτικών μας, είναι δομική, δομικό ελάττωμα της δημοκρατίας μας. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο ε, τμήμα των, του πληθυσμού που δεν εκπροσωπείται. Αυτό σημαίνει ότι τα μόνα τεχνικά όρια, τα μόνα εργαλεία τα οποία έχουν για την προστασία των δικαιωμάτων τους είναι τα δικαστήρια που, τα, δικαιώματα που τους δίνουν τα, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διάφοροι οργανισμοί προστασίας των ελευθεριών και η συζήτηση για τα, για τα δικαιώματα των μεταναστών είναι πάρα πολύ έντονη σε, όλη την, σε όλο τον δυτικό κόσμο, τον ελεύθερο κόσμο, ακριβώς λόγω της ε, ανυπαρξίας των μεταναστών αυτών από άποψη πολιτική. Όμως, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μετανάστες έχουν πολιτικά δικαιώματα, όπως όλοι μας. Έχουν τα, τις ίδιες θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα όπως όλοι μας. Ε, δεν έχουν βέβαια το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε και δεν μπορούν να μπουν σε άλλα κράτη. Ακόμα και το δικαίωμα στην ισότητα και η απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης που σχετίζεται με την ε, εθνική προέλευση. Όλα αυτά τα δικαιώματα τα έχουν οι μετανάστες, όπως όλοι μας. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό από τις κρατικές αρχές και θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα δικαστήρια, από τους, ε, θεσμούς ε, εθνικό, τους εθνικούς προστασίας ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό όμως το ξεχνάμε στην πολιτική συζήτηση που έχουμε πολύ συχνά. Επομένως, αυτό το οποίο τονίζω σαν πρόβλημα είναι η, συχνά η απουσία μιας, ενός κοινού πλαισίου, νομικού πλαισίου για τους μετανάστες. Μου έκανε εντύπωση στις επισκέψεις μου το πώς ε, τα κράτα, κέντρα κράτησης ε, διοικούνται με πολύ με τελείως διαφορετικό τρόπο σε ένα μέρος της χώρας από ένα άλλο. Α δούμε τις φυλακές. Οι φυλακές ακολουθούν ένα εθνικό πλαίσιο, έναν ε, τρόπο, υπάρχει ένα σύστημα εθνικό για τον τρόπο που πρέπει να ε, διοικούνται Δηλαδή, η ποινική κρατούμενη ε, ρυθμίζεται για τον τρόπο με τον οποίο θα έχουν πρόσβαση στην οικογένειά τους, στους δικηγόρους τους, ε, ε, πώς θα τα τρέφονται, πόσες ε, ώρες ελευθερίας ε, θα έχουν ε, ή ε, ε, πόσο πρέπει να είναι το κελί, οι του κελιού τους ή της αυλής τέλο πάντων που θα αυλίζονται κτλ. Η μετανάγκες του μετανάστες δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μια, μια ερώτηση για τα κέντρα κράτηση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στην Ελλάδα που επισκέφθηκα 11 κέντρα ε, και ένα ήταν τραγικό. Και το συζήτησα με τον διευθυντή του κέντρου Κράτηση και μου είπε ότι δύο χρόνια δύο χρόνια μου ζητάω να το κλείσουν και όντως τώρα όντως έχει κλείσει. Μετά όμως την επίσκεψή μας. Όταν εγώ την, όταν εγώ την επισκέφθηκα, και αυτό το κέντρο το, συζητήσαμε στην επιτροπή, στην επιτροπή μας και είπαμε θα το κλείσουμε και έκλεισε. Γιατί το αναφέρουμε τώρα. Λοιπόν, λοιπόν αυτό που είπα όμως ότι, ότι όταν εγώ το επισκέφθηκα ήταν ανοιχτό και έκλεισε μετά. Δεν λέω ότι ήταν σαν συνέπεια τη επίσκεψή μου, εγώ λέω ότι ήταν ανοιχτό όμω και λειτουργούσε όταν ήμουν εκεί. Και προφανώ στην Ελλάδα, στην Ιταλία και σε άλλε ακόμα χώρε. δεν υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε του μετανάστες. Είχα πολύ καλέ εμπειρίε σε άλλα κέντρα κράτηση και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ένα κέντρο κράτηση στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, οι μετανάστες Ε, έχουν, ε, δικούς, έχουν ε, κάποιους χώρους όπου μπορούν να συναντιόνται με τους, με τους συνηγόρους τους, με την οικογένειά τους. Δεν έχουμε συγκρούσεις, είναι πολύ πιο... Ε, δεν έχουμε καμία σύγκρουση και δεν έχουμε διαφορές. Σε, άλλες, σε άλλα κέντρα αυτό δεν επιτρεπόταν ε, και μας είπανε για λόγους ε, ασφάλειας. Τώρα στο κέντρο που τους επέτρεψαν να που επιτρεπόταν να έχουν αυτές τις επαφές μας έλεγαν ίσα ίσα για λόγους ασφαλείας το επιτρέπουμε αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει σε κάθε χώρα να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα με την ε, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, έτσι ώστε να υπάρχει ένας λογικός κατάλογος ε, με τις διατάξεις αντιμετώπισης και συμπεριφοράς απέναντι στους μετανάστες. Λοιπόν, αυτό το οποίο επίσης ε, τώρα ήθελα να πω, ότι ε, τοποθετούμε τους μετανάστες σε μια, σε μια μεγάλη κατηγορία όλους μαζί σαν σακί. Όμως δεν ισχύει αυτό. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι, άρα θα πρέπει να ε, αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα πρέπει να κρατώνται. Πρέπει να τους υποστηρίζουμε, να έχουν πρόσβαση σε ειδικέ διαδικασίες. Η πιστεύω ότι θα στο, στο άμεσο μέλλον θα λειτουργήσει ε, και θα αναλάβει δράση. Αλλά το χρειαζόμαστε αυτά. Επίσης τα παιδιά έχουν ιδιαίτερα δικαιώματα. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να κρατώνται. Αυτή η κράτηση δεν μπορεί να θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον των παιδιών. είδα τα παιδιά πώς κρατώνται τα παιδιά δεν πρέπει να κρατώνται, πρέπει να είναι ελεύθερα. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο, εάν είναι σε ηλικία που ε, πηγαίνουν σχολείο. Αυτό το λέει και ο χάρτης θεμελιωδιών δικαιωμάτων των παιδιών. Οικογένειες με παιδιά δεν θα πρέπει να κρατώνται, γιατί και τα παιδιά δεν πρέπει να κρατώνται και αν μιλάμε για οικογενειακή ενότητα, ούτε και η οικογένεια πρέπει να κρατείται τα άτομα τα οποία έχουν προβλήματα σωματικής ή πνευματικής υγείας. Πρέπει να περιθάλτονται. Και αυτό το οποίο είδα για τα κέντρα κράτηση, αλλά ακόμα και αυτούς που είναι άστεγοι. Δεν έχουν καμία εύκολη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ε, για να μην μιλήσω και για την πνευματική υγεία. Υπάρχουν κάποια προγράμματα, ελάχιστα, κυρίως είναι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, που προσφέρουν ε, υπηρεσίες ε, είτε στο δρόμο είτε στα κέντρα κράτησης, διότι εκεί, που θα, εκεί δεν προβλέπονται ε, τέτοιου, είδη, τέτοιου είδους κανόνες. Κανονικά όμως όταν μιλάμε για κέντρα κράτηση πρέπει να υπάρχουν κάποιες δομές, ε, όπως και στις φυλακές παραδείγματος χάρη. Επομένως υπάρχουν κάποιες ανάγκες τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιήσουμε. Επίσης το, ο στόχος της κράτησης πρέπει να αναφέρεται και αυτό αναφέρεται και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Τον, θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία χαιρόμαστε όλοι μας. Η κράτηση πρέπει να είναι μια τελική, το το τελικό, ε, η τελική δυνατότητα που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας. Και υπάρχουν, ε, και υπάρχουν ε, προβλέπονται κάποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις. Ας πούμε σε κάποιες χώρες έχουν τα ηλεκτρονικά βραχιόλια, α, κάποιοι άλλοι έχουν κάποιους, προβλέπονται κάποιοι εγγυητές αν θέλετε. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κάποια καταφύγια πρέπει, υπάρχουν ήδη καταφύγια για κάποια παιδιά. Οι οικογένειες ε, θα πρέπει να φροντίζονται από τις ε, κοινωνικές υπηρεσίες όλοι οι μετανάστες έχουν διαφορετικές ανάγκες, έχουν θεμελιώδη δικαιώματα και άρα πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι σαν μια ενιαία κατηγορία παρανόμων ή εγκληματιών, θα πρέπει να γίνεται διάκριση και να αντιμετωπίζονται από τις διάφορες υπηρεσίες τις οποίες έχουμε δημιουργήσει για μας. Και σε γενικές γραμμές κάτι το οποίο λείπει ε, γενικά είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Πραγματική και ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Πρόσβαση στην δυνατότητα να, αναθεωρούνται ε, εντολές για απέλαση, για, για επιστροφή και στις χώρες που επισκέφτηκα αυτή η προσφυγή ε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μπορεί να προβλέπεται από τον νόμο, αλλά είναι είναι πάρα πολύ δύσκολη στην Ιταλία. Πρέπει να κάνεις δύο διαφορετικές προσφυγές για την διαδικασία κράτηση και για τη διαδικασία απέλασης και πολλές φορές σε διαφορετικές πόλεις, άρα πρέπει να προσλάβεις δύο διαφορετικούς ε, δικηγόρους. Και μιλάμε για άτομα τα οποία ούτως ή άλλως τον έναν δικηγόρο δεν μπορούν να προσλάβουν. Άρα πρέπει να έχουμε ουσιαστική προσφυγή στην δικαιοσύνη, να υποστηρίξουμε επίσης ε, ε, τους εθνικούς οργανισμούς, τους εθνικούς φορείς, έτσι ώστε να μπορούν να επισκέπτονται τα άτομα αυτά και να ε, αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν τα παιδιά, οι οικογένειες, ε, ασθενείς, ε, ηλικιωμένοι. Ε, έχουν συγκεκριμένες και ειδικέ ανάγκες και αν δεν μπορούν οι κοινωνικέ υπηρεσίε ή μη κυβερνητικέ οργανώσεις να επισκεφτούν τα κέντρα κράτησης, δεν θα γίνει τίποτα. Είδα τραγικές περιπτώσεις στα κέντρα κράτησης. Μία τελευταία παρατήρηση πριν προχωρήσω στην συνέχεια που θα δοθεί σε αυτή την έκθεση. Όχι, όχι, όχι. Ας πάμε κατευθείαν στη συνέχεια που θα δοθεί. Ε, γιατί ε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Στο, στα Ηνωμένα Έθνη, λαμβάνοντας υπόψη τον, ε, τα όρια που υπάρχουν στις ειδικέ διαδικασίες, και εγώ είμαι μια ειδική διαδικασία, είμαι ειδική ομα, όπως οι ειδικές ομάδες, ειδικοί εισηγητές κτλ. Σπάνια επαναλαμβάνουμε την επίσκεψη διότι ας πούμε πρέπει να ασχολούμεθα με 194 χώρες στον κόσμο και σπάνια μας δίνει τη δυνατότητα να επισκεφθούμε ξανά, επισκεφτούμε ξανά μια χώρα. Αυτό το όμως είναι ενδιαφέρον στην διαδικασία του ΟΗΕ είναι ότι η έκθεση αυτή θα προσθεθεί στις εκθέσεις των άλλων ειδικών απεσταλμένων, ε, θα προσθεθεί ε, στις συνθήκες, ε, υπάρχουν και στις στα πρακτικά, αν θέλετε, όλων των ε, επιτροπών που ασχολούνται και θα προσθεθεί και στην ε, περιοδική έκθεση που ε, δημοσιεύεται. Άρα εγώ προσθέτω, σαν ειδικό εισηγητής, προσθέτω γνώση και πληροφορία η, η δουλειά πρέπει να γίνεται από εσά, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, από άλλα κράτη που συζητούν ε, με τις ε, κυβερνήσεις και από τις επιτροπές που συζητούν με τις κυβερνήσεις ε, όταν οι κυβερνήσεις παρουσιάζουν περιοδικές τους εκθέσεις. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον και το οποίο αναφέρθηκε είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά, το να αποδειχθώ λάθος, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν φορέας είναι αντικείμενο ελέγχου από, την, από μια ειδική διαδικασία του ΟΗΕ. Αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Και είναι και ενδιαφέρον διότι αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο έχει έναν ρόλο να παίξει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όχι μόνο έχει έναν ρόλο, αλλά έχει και τεράστια παράδοση ε, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, η Ευρώπη εφήβρε, αν θέλετε, την ομολογία για την ε, ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό το οποίο κάνω τώρα είναι να σας απευθύνω μία έκκληση να διατηρήσετε αυτή την παράδοση όταν αντιμετωπίζετε τους μετανάστες και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε τους μετανάστες δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα θέλετε και τα παιδιά σας να αντιμετωπίζονται στην περίπτωση που γίνουν και αυτά μετανάστες. Σας ευχαριστώ. Ήταν ε, πάρα πολύ ισχυρό το μήνυμα που περάσατε σε αυτή την πρόταση την τελευταία αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για επιμέρους χώρες, αλλά πρόκειται εδώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση το σύνολό της. Σας ευχαριστώ και πάλι και ελπίζουμε ότι θα συνεχίζετε να μας παρουσιάζετε τέτοιου είδου εκθέσεις. Παρακαλώ. Καθίστε, θα συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το 17 έχει αναβληθεί. Okay, <laughs> uh, point which is the Το, η αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναβληθεί. Το επόμενο σημείο είναι η πανευρωπαϊκή έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με τις εμπειρίες εγκλημάτων μίσους και διακρίσεων κατά των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανσεξουαλικών. Θα ήθελα να, ζητή, να παρακαλέσω αυτούς που φεύγουν που εγκαταλείπουν την αίθουσα να το κάνουν ήσυχα. Γιατί συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξή μας. Και αυτοί που θέλουν να παραμείνουν να καθίσουν παρακαλώ. Ούτως ώστε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Πριν ε, ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω ότι στις 17 Μαΐου ήταν ε, η Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας και της τρονσφο τρανσφοβίας. Μελετήθηκε η έρευνα από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αυτών των ατόμων και σήμερα είναι ο Ντένις Βάντερβερ ο οποίος είναι αρμόδιος για την ισότητα των πολιτών, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την παρουσίαση του οργανισμού. Και σας δίνω το λόγο. Εμείς θα φύγουμε από το κέντρο για να βλέπετε τις διαφάνειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την ε, πρόσκληση του Οργανισμού Θεμελιδών Δικαιωμάτων σε αυτή τη συνάντηση για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης έκθεσης για αυτά, αυτή την εμπειρία εγκλημάτων μίσους και διακρίσεων των LGBT ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία. Αυτή η έκθεση ακολουθήθηκε από πολλές ε, κλήσεις και πολλά δεδομένα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων. Πριν παρουσιάσω τα αποτελέσματα και πριν ε, σας δείξω και ένα σύντομο βίντεο για αποτελέσματα αυτά, θα ήθελα να σας ε, διευκρινίσω ότι ο οργανισμός μας έκανε σημαντική εργασία, νομική συγκριτική ανάλυση στην κατάσταση των ΛΟΑΦ ατόμων και κάναμε έρευνες για αυτές τις εμπειρίες ε, διακρίσεων. Αλλά η μελέτη αυτή καθ' αυτή είναι μια τρίτη φάση. Η, ε, έρευνα... είχε, έγινε σε 93.000 άτομα και καλύφθηκαν όλες οι χώρες μπόρεσαν να απαντήσουν τα άτομα στις, ε, στη δική τους γλώσσα και θα σας δώσω ένα σύντομο βίντεο το οποίο θα σας ε, κάνει μια σύντομη εισαγωγή στα αποτελέσματα και στη συνέχεια θα κάνω μια μεγαλύτερη ε, παρουσίαση και θα συνεχίσει η συζήτηση.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 While waiting... Ωραία. Καθώς περιμένουμε θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση, αλλιώς θα χάσουμε όλο το χρόνο. Ήταν η πρώτη, όπως σας είπα, έρευνα αυτού του τύπου που έχει γίνει και βεβαίως η έρευνα ε, ζήτησε ε, να ερευνήσει τις διακρίσεις και τη θυματοποίηση αυτών των ατόμων και βασίζεται σε, στην πολύ, πολύ καλή εργασία που έχει γίνει από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, πληροφορηθήκαμε για το κοινοτικό κεκτημένο, αλλά επίσης και την εργασία των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, ε, ε ιδιαίτερα τη σύσταση 2015. Ε, όπως σας είπα, συμμετείχαν 92.000 στην έρευνα αυτή και καθώς θα δείτε στα αποτελέσματα ενώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 28 χωρών που καλύφθηκαν. Επίσης έχουμε ορισμένα ευρήματα που βλέπουμε ότι υπάρχουν λίγες διαφορές αναχώρα, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκπαίδευση και ε, την κοινωνική πραγματικότητα. Αλλά θα επανέλθω στο σημείο αυτό. Επίσης είδαμε, εξετάζοντας ε, τις νεότερες και μεγαλύτερες ηλικίε ότι οι νεότεροι αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκπαίδευση και την αποδοχή βάσης της ταυτότητας του φύλου.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 αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε τα δεδομένα στη δική μας ιστοσελίδα. Μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα, να δείτε τα αποτελέσματα και να κάνετε τις δικές σας εκτιμήσεις εφόσον επιθυμείτε. Ε, και μπορεί να γίνει ένας διαχωρισμός στις διάφορες ε, υπομάδες ή ανά ηλικιακή κατηγορία, εισοδήματα κλπ. Αλλά ας δούμε πιο προσεκτικά τα αποτελέσματα και θα φωτίσω ορισμένους τομείς, απασχόληση, εκπαίδευση, κοινωνικές πραγματικότητες και επίσης τον τομέα της βίας και των εγκλημάτων μίσους. Ε, ένας από τους λίγους τομείς όπου έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία όταν το θέμα είναι οι διακρίσεις ε, σε σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό είναι ο τομέας της απασχόλησης. Ε, και εδώ ε, ρωτήσαμε τους ερωτώμενους κατά πόσο έγιναν εις βάρος τους διακρίσεις τους τελευταίους 11 μήνες στο χώρο εργασίας τους, ή ζητώντας να προσληφθούν. Και λόγω ακριβώς ότι είναι, ανήκουν σε αυτή την ομάδα. 20% των ερωτηθέτων απάντησαν ότι αισθάνθηκαν να γίνονται εις βάρος τους διακρίσεις. Αισθάνθηκαν ε, να γίνονται διακρίσεις. Ήταν υποκειμενική εμπειρία των διακρίσεων. Όταν δούμε τα αποτελέσματα πιο προσεκτικά διαπιστώνουμε κάτι άλλο. Ότι η, η τρανσεξουαλική ε, αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά διακρίσεων. Και αυτό το έχουμε ακούσει πολύ συχνά από μη κυβερνητικού οργανισμούς. Φαίνεται ότι τα προβλήματα των τασεξουαλικών είναι πιο σοβαρά. Όταν δούμε τι γίνεται στο χώρο εργασίας και βλέπουμε ότι 44% δέχτηκαν αρνητικά σχόλια στην ε, εργασία τους οι 67% άκουσαν τουλάχιστον ένα αρνητικό σχόλιο από κάποιον ε, συνάδελφο. Ε, βεβαίως, σημαντικό είναι να εφαρμόζεται την νομοθεσία και να υπάρχει γνώση του νόμου και να μπορούν ε, τα θύματα να προσφεύγουν στο νόμο. Ε, ζητήσαμε να υπάρξει σχετική νομοθεσία που να απαγορεύει ε, τις διακρίσεις. Ε, ε, και συγκρίναμε τα στοιχεία αυτά με τις νομοθεσίες προστασίας των μειονοτήτων. Επίγνωση του νόμου είναι 84% το ποσοστό στη Σουηδία, αλλά μόνο 21% είναι η γνώση του νόμου στην Κύπρο. 10% όσων ανέφεραν ότι αισθάνονται διακρίσεις βάρες τους στο χώρο εργασίας και το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό εν σχέση με τις άλλες ε, ομάδες που γίνονται θύματα διακρίσεων. Ε, το 90% δηλαδή δεν αναφέρουν αυτές τις διακρίσεις εναντίον τους. Και εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των χωρών μελών, μπορούμε να τα δούμε στην οθόνη. Βεβαίως η απασχόληση δεν είναι ο μόνος ε, τομέας όπου γίνονται διακρίσεις. Εξετάσαμε άλλους τομείς πέραν της ε, εργασίας, τομείς ε, που καλύπτονται από την πρόταση οριζόντιας οδηγία. Εξετάσαμε για παράδειγμα τι γίνεται στην εκπαίδευση, στη στέγαση, στι υπηρεσίε υγεία, αλλά επίσης όταν κανείς πηγαίνει σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπάρι, σε ένα κατάστημα, κατά πόσο βιώνει διακρίσει ε, εναντίον του σε αυτούς τους χώρους και εκεί βρήκαμε ότι 32% κατά μέσο όρο για όλες τις ηλιακέ ομάδες ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν κάποιες διακρίσεις βάρος τους τους 20 μήνες πριν από την διεξαγωγή της έρευνας. Και πάλι υπάρχουν εδώ διαφορές αναχώρα και αναομάδα. Οι λεσβίες και οι τρανσεξουαλικοί ε, βρίσκονται στα δύο άκρα. Ε, στο τέλος της ε, έρευνας αφήσαμε ανοιχτή τη δυνατότητα να κάνουν κάποια σχόλια και 23.000 από τους ερωτηθέντες ε, σχολίασαν ε, μακροτενώς την εποχή για παράδειγμα που πήγαιναν στο σχολείο και τις διακρίσεις που είχαν υποστεί λόγω του προσανατολισμού του φίλου και το πώς είχαν αισθανθεί οι ίδιοι μαθητές. Στον τομέα της εκπαίδευσης, αυτός είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου βρήκαμε πραγματικά εντυπωσιακέ ομοιότητες μεταξύ των χωρών. Όταν ρωτήσαμε τους ερωτηθέντες κατά πόσο είχαν ακούσει αρνητικά σχόλια ή είχαν αρνητικές εμπειρίες από του συμμαθητές τους, ε, διαπιστώσαμε σε όλες τις χώρες μέλη μέχρι από 83% σε 97% και πολύ λίγες διαφορές ε, μεταξύ των υποομάδων λεσβιών, ομοφοφίλων, αμφισεξουαλικών κλπ. Ε, άρα φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα ε, και επίσης ρωτήσαμε κατά πόσο ξεσκέπασαν την ταυτότητά τους ε, κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ηλικίας. Ε, και εδώ υπάρχουν πολύ λίγες διαφορές. Ε, ένας μέσος αναχώρες, 67% είναι ο μέσος όρος και είναι ενδιαφέρον ότι μπορούμε να δούμε ιδιαίτερα όσον αφορά την, τους τρανσεξουαλικούς τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά. Τώρα, Επίσης επικεντρώσαμε την προσοχή μας σε περιστατικά βίας, εγκλήματα μίσους και ευρύτερα ε, πού βλέπουν οι άνθρωποι αυτοί ένα ασφαλές περιβάλλον και κατά πόσο αισθάνονται ασφαλείς όταν βγαίνουν στον δρόμο, πηγαίνουν κάπου κλπ. Και τους ρωτήσαμε τον ίδιο τρόπο όπως το κάναμε σε σχέση με άλλε ομάδε που να διακρίσει ε, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν, ε, τους ρωτήσαμε κατά πόσο είχαν εμπειρία βία τα τελευταία πέντε έτη ή και κατά πόσο είχαν εμπειρία βία τον τελευταίο χρόνο. Για τα πέντε χρόνια ήρθαμε στο ποστό 26% για κατά 26% είχαν υποστεί σωματική βία ε, και πάλι εδώ οι τρανσεξουαλικοί αναφέρουν ένα 35% ιδιαίτερο υψηλό ποσοστό εντός της ομάδας. Για τους τελευταίους 12 μήνες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 10%. Και πάλι εάν δούμε κατά πόσο αναφέρουν οι άνθρωποι αυτά τα περιστατικά στην αστυνομία, βρήκαμε ότι μόνο 22% όσων είχαν βιώσει βίο περιστατικό το ανέφεραν στην αστυνομία. Και πάλι πολύ χαμηλό το επίπεδο. Ο λόγος για τον οποίο δεν αναφέρουν αυτά τα περιστατικά ε, βίας είναι ότι δεν εμπιστεύω την αστυνομία, δεν θα αλλάξει τίποτα, καμιά φορά δεν ξέρουν που να αποτανθούν και υπάρχουν και κάποια θέματα ε, ε, ε, άρα υπάρχουν κάποια θέματα με τα οποία θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Ε, όταν δούμε λοιπόν αυτό το 10% που ανέφεραν περιστατικά βία το τελευταίο έτος, 59% των όσων είχαν δεχτεί επίθεση απόδωσαν την επίθεση στην ταυτότητα φίλου, του σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Και πάλι εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Ο τελευταίος τομέας και βεβαίως ε, μπορώ να επιλέξω μόνο μερικά στοιχεία από την παρουσίαση είναι αυτό που ονομάζουμε καθημερινή ζωή και κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή πώς βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί τα θεμελιώδη του δικαιώματα σε καθημερινό επίπεδο, όταν βγαίνουν στον δρόμο, όταν πάνε στο σχολείο, αλλά επίση στο σπίτι του και στο εγγύ του περιβάλλον. Ένα ερώτημα το οποίο θέσαμε είναι κατά πόσο ε, κρατιούνται χέρι-χέρι με τον αγαπημένο του ή τον σύντροφό του στον δρόμο. Και οι εκριβής ερώτηση κατά πόσο αποφεύγουν να πηγαίνουν χέρι-χέρι σε δημόσιο χώρο. Και είδαμε τα αποτελέσματα όπου κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση στην Ισπανία και την Δανία, όπου οι άνθρωποι αναφέρουν χαμηλότερα ποσοστά αποφυγής και 89% είναι στην Κροατία και την ε, Κύπρο επί παραδείγματι. Άρα λοιπόν οι ομοφιλόφιλοι άνδρες αποφεύγουν να κρατούνται από το χέρι δημοσίως. Ε, και αυτά τα αποτελέσματα και πολλά άλλα βεβαίως ε, χρήζουν κατάλληλης ε, απόκρισης, αντίδραση. Και καταρχήν ρωτήσαμε του ρωτηθέντε, τι πιστεύουν θα πρέπει να γίνει για να βελτιωθούν τα δικαιώματά τους Και στην οθόνη μπορείτε να δείτε μερικές από τι απαντήσει που δόθηκαν πολύ συχνά. Για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να βελτιωθούν, να εφαρμοστούν κάποια μέτρα στο σχολείο, να υπάρξει ένα περιβάλλον ασφαλές από bullying, ε, επίσης να υπάρχει κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων και οι εθνικές ε, αρχές επίσης, να, οι δημόσιες αρχές να, προσπίζουν αυτά, να υπερασπίζονται αυτά τα δικαιώματα. Ε, στην έρευνα είδαμε ότι οι ερωτηθέντες ε, γνωρίζουν ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες από τις ε, κυβερνήσεις, από τις χώρες και ε, σε εκείνες τις χώρες όπου γίνεται η προσπάθεια να ληφθούν κάποια μέτρα, αυτό όντως εμέσως συνάγεται από την έρευνα, βιώνεται θετικά από τους ερωτηθέντες. Και βεβαίως ε, εμείς διατυπώσαμε και τις δικές μας ε, απόψεις και συστάσεις προς τις ε, ευρωπαϊκές χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη. Καταρχήν είπαμε ότι αν υπάρχουν προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κροατία και χρειάζονται αντιδράσεις σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο ε, χρειάζονται νομοθετικές αλλαγές για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ο προσανατολισμός του φύλου και η ταυτότητα του φύλου θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητά στην νομοθεσία κατάργηση των διακρίσεων ε, και θα πρέπει να γίνεται ρητή η επισήμανση και διευκρίνηση στον Ευρωπαϊκό Νόμο. Όσον αφορά τώρα τα αποτελέσματα ε, για την εμπειρία των διακρίσεων πέραν ε, της, ε, του χώρου εργασίας είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει ανάγκη νομοθεσίας, ευρωπαϊκής νομοθεσίας που να αφορά και άλλους χώρους πλην του χώρου εργασίας. Τέλος, όσον αφορά τα εγκλήματα βίας και μίσους, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η ομοφοβία και η φοβία έναντι των τρανσεξουαλικών ατόμων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επίσης και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Όπως σας είπα, ε, στην αρχή είχαμε μια πραγματικά, είχαμε πραγματικά ένα πολύ καλό διαλογικό online εργαλείο και μπορείτε να βρείτε όλες τις ερωτήσεις της έρευνάς μας, μπορείτε να δείτε ποια είναι ακριβώς τα αποτελέσματα αναχώρα και βάσει άλλων μεταβλητών. Είναι μια πραγματικά μοναδική πληροφορία που μπορεί να έχουν οι ευρωπαϊκοί φορείς και όσοι χαράσουν τη σχετική πολιτική ε, για την πραγματικότητα αυτών των ανθρώπων. Δεν εξήγησαν πολλά πράγματα σχέση με τη μεθοδολογία. Ε, αναφέρομαι σε αυτό διότι όντως υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε σχέση με όλες αυτές τις μεγάλες ε, επιγραμμικές ε, δημοσκοπήσεις όπου όλοι εκφράζουν την αποψή του ανώνυμα και μετά από πολλές διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και τους, τη δική μα επιστημονική επιτροπή καταλήξαμε στο ότι ο στόχος να καλύψουμε την πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή των ΛΟΑΦ ακόμη και αυτών που δεν το έχουν παραδεχθεί γενικότερα στον κόσμο ή δεν έχουν αποκαλύψει αυτή τη σεξουαλική του προτίμηση στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον ή γενικότερα και θέλουμε ε, στην Ήπεθρο, στη Ρουμανία να καλύψουμε παραδείγματο χάρη της ε, λεσβείε ε, ή στη, στο City του Λονδίνου έναν μορφωμένο νεαρό. Ε, υπήρχε επικοινομορφία δηλαδή στους ερωτηθέντες και έχουμε χρησιμοποιήσει διάφορες παραμέτρους για να καλύψουμε διαφορετικά προφίλ ερωτηθέντων. Ε, σύντομα θα έχουμε ε, περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα για σας ε, στον ιστότοπό μας αφού θα έχουμε αναλύσει περαιτέρω τα πορίσματα της μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much uh, for the report. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Πριν από εσά ήταν εδώ ο εκπρόσωπο ε, τη ΥΠΑ τη Αρμοστία του ΟΗΕ που μα κυαγράφησε μια όχι τόσο πολλά υποσχόμενη κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω έχουμε πολλά να μάθουμε σε σχέση με το ε, πώ πρέπει να προχωρήσουμε για αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα. Έχουμε τώρα χρόνο για ερωταπαντήσει, παρατηρήσει, συζήτηση. Ποιο θα ήθελε το λόγο. Μπίργκετ Σίπερ θα πάρει πρώτα το λόγο και μετά θα ακούσουμε τα υπόλοιπα σχόλια. Ε, ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώ, ε, δεν ήμουν παρούσα σε όλη τη διάρκεια τη παρουσίαση. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο το οποίο θεωρώ ιδιαίτερο σημαντικό. Στην έκθεσή σα εξετάσατε τι πιστεύουν οι ίδιοι ερωτηθέντε ότι θα πρέπει να γίνει προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Και πολύ ψηλά στη λίστα ήταν το ότι θα πρέπει άτομα που έχουν θρησκευτικά αξιώματα και πολιτικοί να δηλώσουν δημοσίως ότι είναι υπέρ των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Και πραγματικά είναι σχετικό το γεγονός ότι αυτές τις μέρες ε, γίνονται, γίνεται ακριβώς το αντίθετο εκ μέρους των πολιτικών προσώπων ή θρησκευτικών φορέων. Και αυτό πραγματικά είναι ανησυχητικό και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν εμείς από το ευρωπαϊκό επίπεδο να αποστείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Ε, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα όταν σε εθνικό επίπεδο ε, γίνονται εκ των άνω ε, διακρίσεις εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Νομίζω ότι θα πρέπει εμείς τουλάχιστον να καταγγέλουμε αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγορητή για την παρουσίαση. Θέλω να κάνω κάποιους παραλληλισμούς. Το θέμα της ε, νομοθετικής δράσης κατά τη διαστολή με το θέμα της παιδείας ε, και της ε, κατανόησης είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία και σε άλλους τομείς. Εγώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είχα αναλάβει τη δεκαετία του 90 την διοίκηση μιας σχετικής υπηρεσίας και ήταν πολύ λεπτή ισορροπία ακριβώς ε, ανάμεσα στην νομοθετική προσέγγιση, της υποχρεωτικέ διατάξεις αφενός και αφετέρου ότι να βρούμε τη σωστή προσέγγιση για να έχουμε και την καλή διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση όλων για τέτοια ζητήματα. Ε, η διακριτική μεταχείριση, φιλετική ή άλλη, συχνά ε, απηχείται και σε διάφορα πολιτικά φρονήματα ε, ή έρχεται ως απόρρια άλλου είδους πίεσης ε, που ε, ασκείται σε κάποιους. Κάποιοι δηλαδή αντιλαμβάνονται αυτό ως καταπίεση, ως ένα είδος πίεσης. Είναι κάτι απαράδεκτο και όντως χρειάζεται πολύ αυστηρή στάση από πλευράς ε, κάθε κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε ένα ορισμένο βαθμό, όμως είναι δύσκολο να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Και επίση θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το ποιο βαθμό λεπτομέρειε επιδιώκουμε στην ε, παρασκευαστική μα ε, άσκηση, γιατί μπορεί να έχουμε και το αντίστροφο αποτέλεσμα να ενισχύσουμε αυτή τη διακριτική μεταχείριση. Ε, αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε στην ε, ε διαπαιδαγώγηση, στην ε, συμφιλίωση για να μας ακολουθήσουν ε, οι πολίτες και να ελεγχιστοποιήσουμε τις περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης. Εγώ πιστεύω πως είναι απαράδεκτη κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης, όμως εξίσου σημαντικό είναι να είμαστε λογικοί και ρεαλιστές στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα ε, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όλοι όσοι έχουν βρεθεί σε κατάσταση μειονότητας για οποιοδήποτε λόγο. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ χρήσιμα τα στοιχεία για τη σημερινή μας συζήτηση. Ευχαριστούμε, λέει η Προεδρεύουσα είναι σημαντικό να δούμε και τι συμβαίνει στα σχολεία και από αυτή την πλευρά έχετε δίκιο. Η παιδεία είναι ένα στοιχείο κλειδί πέρα από αυτούς που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, το ρόλο των πολιτικών, τη νομοθεσία. Η κυρία Λούνατσεκ θα πάρει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ αρχικά να ευχαριστήσω την Υπηρεσία Θημελιωδιών Δικαιωμάτων που ε, έκανε την ε, δημοσκόπηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο είχαν ζητήσει να διεξαχθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα για μας. Πρώτη φορά έχουμε μια επισκόπηση ε, για την καθημερινή ζωή, φόβους, ανησυχίες και διακριτική μεταχείριση που βιώνει η ΛΟΑΦ. Ε, είναι η πρώτη φορά εγώ ε, είμαι λεσβία εδώ και 30 χρόνια και εδώ και 20 χρόνια ε, είμαι στην πολιτική. Ε, και και έχω ασχοληθεί επισταμένα με αυτό το ζήτημα. Ήμουνα στη Χάγη πριν από δύο εβδομάδες με διάφορους βουλευτές και άκουσα την παρουσίαση στις 17 Μαΐου που ήταν η Διεθνής ημέρα των ΛΟΑΦ. η πρώτη αντίδραση μου ήταν επίσης ότι το, ο φόβος, το μέγεθος του φόβου που αποκαλύπτεται όταν μαθαίνουμε τις λεπτομέρειες καθημερινής ζωής αυτών των ανθρώπων είναι κάτι τρομακτικό και για μας. Εγώ δεν πιέζω συνήθως για να συζητάμε για τα κακό κείμενα. Εγώ προσπαθώ αντίθετα να δίνω θετικά παραδείγματα ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν χωρίς φόβο, πιο ελεύθερο. Όχι μόνο η ΛΟΑΦ και άλλες κατηγορίες πληθυσμιακέ. Ε, και στη Χάγη όταν με ρώτησαν ε, δημοσιογράφοι δεν είναι, ε, τρομακτικό, δεν είναι τρομακτικά αυτά τα στοιχεία. Συμφώνησα, αλλά είναι η πρώτη φορά που τα μαθαίνουμε. Ας το αναγνωρίσουμε λοιπόν και ας διαπιστώσουμε πόσο διάχυτος είναι ο φόβος. Παρόλη αυτή την νομοθεσία που έχουμε, παρότι έχουμε σε όλες τις σφαίρες της δημόσιας ζωής, στην πολιτική, στην καλλιτεχνική ζωή, στις επιχειρήσεις, σε πολλούς ΛΟΑΒ σε σχέση με το παρελθόν έχουμε και περισσότερα στοιχεία γι' αυτό, αλλά ε, είναι τρομακτικό το να διαπιστώνουμε πόσο διάχυτος είναι ο φόβος. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποιες διαστάσεις του Δήμους που θίξατε και εσείς και ο κύριος Κύρκοφ. Είπατε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά σχόλια στον εργασιακό χώρο, στα σχολεία, στο εκπαιδευτικό σύστημα και νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα της μελέτης ε, για αυτούς που μας λένε δεν πρέπει να δείχνεστε τόσο πολύ, να φαίνεστε τόσο πολύ, να ζητάτε, να προβάλλετε την εικόνα των ΛΟΑΦ διότι ε, ε, ε όμως αυτό χρειάζονται αυτοί που φοβούνται είτε μιλούμε για ε, ΛΟΑΦ είτε ε, για ετερόφιλους ε, θέλουμε υποστήριξη από όλους και θέλουμε να μπορούμε να σχολιάσουμε το ότι χθε στη Γαλλία παραδείγματο χάρη έγινε ο πρώτος γάμος ομοφιλοφίλων παρόλες τις διαμαρτυρίες. Μας δείχνει αυτό ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα θετικά σχόλια, ούτω ώστε να κάνουμε την υπέρβαση και να υπερπηδήσουμε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια που δεχόμαστε. Νομίζω όλοι ε, μπορούμε να το πετύχουμε αυτό στην καθημερινή μα ζωή, στην επαγγελματική και ιδιωτική μα ζωή. Με προσωπική κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση. Κάτι άλλο τώρα για την ε, παιδεία και τη διαπαιδαγώγηση. Είναι κεντρική σημασία. Στο σχολείο μαθαίνουν τα παιδιά όταν είναι πάρα πολύ μικρά τι ε, είναι αποδεκτό και τι δεν είναι. Και ο εκφοβισμός ε, στα σχολεία, το bullying ε, ή κατά τον αθλητισμό έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στον αθλητισμό. Είχα, ήμουνα οπαδός, σε διάφορα αθλήματα και παραδείγματο χάρη στη Γερμανία στο σχολείο μου είπαν ξέρετε πώς αποκαλούν ε, αυτούς τους ανθρώπους γκέι. Ε, δηλαδή κάποια παιδιά, θα το λέω αυτό το παράδειγμα για να καταλάβετε ότι κάποια παιδιά ε, δεν ήξεραν καν τι σημαίνει γκέι ομοφιλόφιλος ε, γιατί θεωρούσαν ότι είναι κακή λέξη και ότι δεν είναι αρκετά άντρας ένας άντρας που είναι ομοφιλόφιλος για να παίξει ποδόσφαιρο παραδείγματο χάρη. Ε, φαίνεται ότι χρειαζόμαστε εγχειρίδια σχολικά, πραγματική διαπαιδαγώγηση που θα προβάλλουν θετική εικόνα για τους ε, ΛΟΑΦ ε, από οικογένειε, ουράνιο τόξο όπως ονομάζονται, οικογένειε δηλαδή ομοφιλοφίλων, ε, οι οποίες όμως υπάρχουν όλα και συχνότερα στην κοινωνία. Πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Οι, δάσκα, οι δάσκαλοι που αποκαλύπτουν τη σεξουαλική τους προτίμηση επίση, άλλο ένα σημαντικό θέμα, αφού τολμούν ε, να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους και δεν φοβούνται να, ε, θεωρεί, ε, δεν φοβούνται να θεωρηθεί παραδείγματος χάρη ότι προσπαθούν να αποπλανήσουν τα παιδιά. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί μια τέτοια συμπεριφορά. Είναι πολυδιάστατο το θέμα. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε κάτι που μας είπε ο κύριος Κύρκοφ, ο συναδελφός. Είπατε ότι η υπερβολικά λεπτομερής νομοθεσία ενδεχομένως και να ενισχύσει τη διακριτική μεταχείριση. Ε, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Πιστεύω ότι σε, σε μια οριζόντια οδηγία κατά της διακριτικής μεταχείρισης ε, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, ε, φιλετικής προέλευση, πολιτικών φρονιμάτων και την το καθεξής, θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες στην νομοθεσία. Για ποιο λόγο, διότι ε, αν δεν υπάρχουν λεπτομερείς ρυθμίσεις ε, δεν τολμούν οι ΛΟΑΦΑ να ε, αποκαλύψουν ταυτότητά τους. Θέλετε να νοικιάσετε ένα διαμέρισμα και φοβάστε ότι ο σπιτρινικοκύρης θα σας αρνηθεί γιατί είστε λεσβία. Άμα το φοβάστε αυτό δεν θα το πείτε. Εάν όμως μπορούν κάποιοι να κάνουν την προσφυγή στην δικαιοσύνη, καταλαβαίνετε πρέπει να κατοχυρωθούν ισότιμα δικαιώματα για όλους. Θα συμφωνήσω όμως μαζί σας ότι κεντρικό ρόλο παίζει η παιδεία. Έχω πολλά να πω, αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσω ζητώντας από κάποιον ή κάποια από την Επιτροπή, δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει, το εξής. Ε, στη Χάγη, αυτό που συνέβη επίσης, και τώρα δεν μιλώ μόνο εξ ονόματος πολιτικής μου ομάδας, αλλά με την ιδιότητα της ε, προέδρου μίας, ε, της συμπροέδρου μάλλον της διαφυλετικής διακομματικής ομάδας για τους ΛΟΑΦ. Ε, ερωτήθη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Χάγη ποια, ποια είναι, ποιες είναι οι προθέσεις για έναν οδικό χάρτη, όπως έχουμε για τους Δρόμα, αλλά για τους ΛΟΑΦ. Ε, η Επίτροπος Ρέντινγκ ακόμη και όταν βρεθήκαμε στη Χάγη δεν ετάχθη πέρα αυτού, δεν υποσχέθηκε ότι θα γίνει αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας. Είπε ότι το δικό της οδικό χάρτη τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολλά πράγματα και έχει σημειωθεί πρώτος, το ξέρουμε και το αναγνωρίζουμε και το εκτιμούμε. Όμως κάτι ε, όπως ένας οδικός χάρτης που δίνει και στα κρατημέλη και στις κυβερνήσεις ένα τρόπο, ένα σημείο αναφοράς ε, με, ώστε ε, ε, ε, οι ψηφοφόροι τους ή όσοι δεν θέλουν να συμμορφωθούν με την νομοθεσία, προώθηση τη εικόνα των ΛΑΦ, ενημερωτικό υλικό και το καθεξής. Θα είναι λοιπόν αυτό το σημείο αναφορά χρήσιμο για όλου και ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Όποιο ε, τελικά θα μα απαντήσει, να μα πει αν κατά τη γνώμη του είσαι, υπάρχει ακόμη η πιθανότητα να συμβεί αυτό. 11 φορέ το έχουμε ζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε, Ουλερή, καλή Προεδρεύουσα. Ε, από όσο ξέρω, Έχουμε κάποιους που εκπροσωπούν εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως ε, θα ήθελα πρώτα να ακούσουμε τους βουλευτές και ε, στη συνέχεια θα ακούσουμε κάποιον ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να μας απαντήσει. Είναι ξεκάθαρη εικόνα και η ερώτηση και χρειαζόμαστε και μια ξεκάθαρη επίσης απάντηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί το Κοινοβούλιο ήταν ξεκάθαρο ζητάμε ε, στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει επιτέλους με την οριζόντια οδηγία για τη διακριτική μεταχείριση ο, ακούσουμε τον κύριο Κλέης πρώτα και μετά ε, τους υπόλοιπους βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ ε, ένα μεγάλο ποσοστό λέει ότι ήταν θύματα ε, σωματικής βίας και αυτό αποτελεί πραγματικό σκάνδαλο. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Στην... Ε, και δεν υπάρχουν και πληροφορίες για τα άτομα τα οποία διέπραξαν τα αδικήματα αυτά το 95% των ε, ε, υπευθύνων για τις σωματικές αυτές επιθέσεις είναι μουσουλμάνοι. Γιατί αυτό το θέμα δεν το αντιμετωπίζουμε και γιατί δεν το ε, συζητάμε καθόλου. Συζητήσαμε για τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη και έγινε και μία αναφορά ε, και στην ε, παρέμβαση των ε, μουσουλμάνων. Αυτό όμως σιωπήθηκε εκ των υστέρων. Εγώ διαφωνώ. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με την λύση, δεν μπορούμε να βρούμε λύση στα προβλήματα εάν δεν ασχοληθούμε και με την προέλευση των προβλημάτων. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και ρωτώ γιατί δεν υπάρχει αναφορά καθόλου στους υπευθύνους των ε, ενεργειών αυτών. Νομίζω ότι είναι λάθος ε, να συμπεριλάβουμε σε μία κατηγορία όλα, την διακριτική μεταχείριση, τις απειλές, ε, την την βία ε, και να μην υπάρχει καμία απόχρωση. Προφανώς κανείς δεν θα πρέπει να ε, αποτελεί αντικείμενο βίας ή απειλών ή οτιδήποτε. Αλλά πού θα φτάσουμε, θα συλλαμβάνουμε ε, ανθρώπους γιατί κάνουν αστεία, θα λέμε στους εκκλησίες, θα στις εκκλησίες και θα λέμε στους ανθρώπους τι πρέπει να πιστεύουν και τι δεν θα πρέπει. Η λεκτική βία και ε, γενικώ αποτελεί κομμάτι του παρελθόντος για, για κάποιες κατηγορίες. Όμως στις μουσουλμανικές ε, περιοχές του Λονδίνου υπάρχουν αφήσεις ε, που προειδοποιούν τους ομοφιλόφιλους να μένουν μακριά και κάποιοι οι οποίοι δεν άκουσαν τις συμβουλές αυτές ε, το πλήρωσαν. Τώρα το πρόβλημα είναι τι γίνεται ε, όταν μία μειονότητα επιτίθεται σε μια άλλη μειονότητα και τις δύο ε, μειονότητες τις υποστηρίζουμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η σεξουαλική προτίμηση κανενός, φίλων, γνωστών, συνεργατών, συναδέλφων κτλ. Δεν με ενδιαφέρουν οι προσωπικές λεπτομέρειες ε, και για τη ζωή των γνωστών μου. Το bullying στα σχολεία, ο εκφοβισμός στα σχολεία πρέπει να απαγορεύεται. Και ο, ο εκφοβισμός ο, ο οποίος... Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι ο εκφοβισμός στα σχολεία είναι μόνο για τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή για τις υποτιθέμενες σεξουαλικές προτιμήσεις ε, των παιδιών. Ο εκφοβισμός πρέπει να σταματήσει Τελεία και παύλα. Διότι τα σχολεία πρέπει να, να μαθαίνουν στα παιδιά ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν τους... Ε, ε, ε, τους ανθρώπους, τους, συνα, τους με κατανόηση και ανοχή και στο σχολείο και ενήλικ και μετά. Κυρία Λούνατσεκ, θα πάρετε το λόγο για άλλη μια φορά, συντομία όμως, και με την πρέπει να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Απλώς ε, θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτά τα οποία είπαν οι δύο συνάδελφοι. Ο κύριος Κλέσα αναφέρθηκε ότι στο 95% των υπευθύνων ε, φαίνεται ότι είναι, εκείνος θεωρεί ότι είναι μουσουλμάνος. Δεν το λέω εγώ, λέει ο κύριος Κλέσα. Εγώ να σας πω ότι είμαι κατά οποιασδήποτε βίας που προέρχεται από οποιονδήποτε. Όμως δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει να εστιάσουμε και να κατηγορήσουμε μία μόνο θρησκευτική ομάδα. Γιατί είδατε και με τις διαμαρτυρίες στην Γαλλία. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο υπήρχαν βία επεισόδια στη Γαλλία και δεν ήταν μουσουλμάνοι, ήταν χριστιανοί. Επομένως, οι φανατικοί, οι φανατικοί από οποιαδήποτε θρησκεία και προέρχονται ή και άθεοι να είναι, αυτοί αποτελούν το πρόβλημα και όχι κάποια θρησκευτική ομάδα και ο κύριος Μπρόνς είπε ότι υπάρχουν οι εκκλησίες ε, και τι θα, λέμε, τι... τι... θα τους πούμε τι θα πιστεύουν. Όχι, εγώ δεν είπα τι θα, θα τους πούμε τι θα πιστεύουν, θα τους λέμε τι θα λένε, διότι δεν μπορούν να πρεσβεύουν ε, το μίσος εναντίον κάποιων ομάδων, γιατί ε, υπάρχει το θέμα τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα όπου υπάρχουν πολλοί διστάμενες απόψεις. Εάν θέλετε να απαντήσετε μπορούμε να το κάνουμε, αλλά μην διακόπτετε τους άλλους. Κύριε Κλής, εν συντομία. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Όλοι όσοι ε, ασκούν βία πρέπει να αντιμετωπίζονται, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Όμως, εάν δείτε ότι το 95 προέρχεται από μία συγκεκριμένη ομάδα, τότε για λόγους αποτελεσματικότητας θα πρέπει να έχεις στο στόχαστρο αυτή την ομάδα για λόγους πρόληψης, αν θέλετε. Η Σόφη θέλει να πάρει το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα αλλά πρέπει να αντιρρήσω σε αυτή την ρατσιστική ανοησία. Κύριε Κλής, όντως δεν υπάρχει καμία θρησκεία που έχει το μονοπόλιο της βίας και της ομοφοβίας και το έχουμε δει παντού. Πάρα πολύ συχνά προέρχεται από οποιαδήποτε θρησκεία. Να μην ακούσω τι λέει το Βατίκανο για, τα, για τις λεσβίες και τους ο, γενικώ και στην Ανατολική Ευρώπη ήρθα σε επαφή με Ορθοδόξους χριστιανούς που ήταν πολύ βίαιοι. Επομένως, όντως συμφωνώ ότι αν δεν ξέρεις την, την ρίζα του προβλήματος δεν μπορείς να το αντιμετωπίσει. Όχι, κλιέσε Έχετε λάθος τα ε, στοιχεία στη διάθεσή σας που έχετε και το να ασκείτε διακριτική αντιμετώπιση ενώ μιας ομάδας δεν βοηθάει και τις υπόλοιπες. Ευχαριστώ θα κλείσουμε τώρα την συζήτηση και θα ήθελα να ακούσω κάποιον από την Κομισιό. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Καλημέρα σας. Λέγομαι Χουάν Γκονθάλες. Ε, ε, δουλεύω στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη στο τμήμα κατά των διακρίσεων και έρχομαι για πρώτη φορά σε αυτή την Επιτροπή. Λυπούμε ότι δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω ή κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είπε, είχε πει η κυρία Ρέντινγκ στο παρελθόν. Αναφερθήκατε στις δράσεις της, Ευρωμένης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και το χάρτι τη χάρτα θεμελιδών δικαιωμάτων και υπενθύμησε στις χώρες μέλη τη μεγάλη τους ε, ευθύνη, την ευθύνη που φέρουν για την ε, πρόθεση των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων και επίσης τόνισε η κυρία Ρέιντινγκ την ανάγκη να θεσπιστεί μια ειδική νομοθεσία προστασίας των ΛΟΑΦΑ και μια σωστή εφαρμογή της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων θα πρέπει να υπάρξει, είπε. Ε, ξέφρασε τη δέσμευση εκ μέρους της Επιτροπής ε, για το θέμα αυτό και εγώ μπορώ να σας ε, διασφαλίσω ότι στην Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης έχουμε αναλάβει μια πλήρη δέσμευση για το θέμα αυτό και θα μπορούσα να σας παρουσιάσω κάποια από τα πράγματα που κάνουμε τους, ε, που θα κάνουμε τους προσεχείς ε, μήνες. Η κυρία Αντιπρόεδρος, η κυρία Ρέντινγκ, είπε ότι υπάρχει στενή συνεργασία με τις χώρες μέλη και παρέχεται οικονομική στήριξη προς αυτές. Ε, υπάρχει η έρευνα σε σχέση με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και μετά το καλοκαίρι θέλουμε να ενώσουμε όλες τις χώρες, να συγκεντρώσουμε όλες τις χώρες που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, να πάρουμε τα αποτελέσματα της ε, έρευνας, ε, την ομοφοβία ή την φοβία ενάντια τρανσεξουαλικών ε, στο σχολείο, το θέμα της εκπαίδευσης κλπ. Ακούσαμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών και υπάρχουν λόγια τους οποίους τα πράγματα δουλεύουν σε κάποιες χώρες και σε άλλες όχι. Και θα μπορούσαμε να προβούμε σε μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τέθηκε στη συζήτηση στο πάνελ εκεί ότι η Κομισιόν θα πρέπει να οργανώσει μια συζήτηση με τις χώρες ε, μέλη γύρω από το θέμα αυτό. Και κάτι το οποίο ήδη κάνουμε, αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη κάνουμε εδώ και τέσσερα χρόνια. Θα ήθελα να σας ε, διασφαλίσω ότι θα υπάρξει μια παρακολούθηση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων και πρόκειται να εθαρρύνουμε τις χώρες μέλη να ενισχύσουν αυτά τα δικαιώματα και ενδεχομένως να χρηματοδοτήσουμε κάποιες εκστρατείες για την καλύτερη επίγνωση των δικαιωμάτων αυτών των μειονοτήτων. Εντείνουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας στον τομέα αυτό και θέλουμε και την συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε το λόγο. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορείτε να πάτε πέρα από ε, τα όρια εκείνων που ήδη είπε η κυρία Ρέντινγκ ε, Αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο μετά από τη διενέργεια αυτής της έρευνας του Οργανισμού Θημελιωδών Δικαιωμάτων ότι κάτι θα πρέπει να γίνει. Ε, σε διάφορους τομείς αναφέρθηκε η οριζόντια οδηγία για τις διακρίσεις αλλά θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα για τα, στον κανονισμό για τα δικαιώματα των πολιτών, να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα αυτών των ομάδων. Και αναφέρεται κάποιες άλλες ε, δράσεις που προγραμματίζεται, αλλά νομίζω ότι υπήρξε κάποια απογοήτευση εδώ στην αίθουσα. Δεν ξέρω αν έχετε επίγνωση αυτής της απογοήτευσης. Ε, και ίσως είναι σημαντικό λοιπόν να καταλήξετε σε κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις από τη δική σας πλευρά, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση και στο επίπεδο των χωρών μελών, να δούμε τι προοπτικές συνεργασίες υπάρχουν. Και τώρα θα ήθελα να σας ζητήσω να πάρετε το λόγο μετά από αυτή την πολύ ζωντανή και ίσως και τόσο, όχι και τόσο εύκολη συζήτηση, να κάνετε ίσως και τα δικά σας σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια σε αυτή την αίθουσα. Έγιναν, ε, υπόθηκαν πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Το πρώτο που αφορά τη σημασία των ε, όσων κατέχουν κάποια θρησκευτικά αξιώματα ή των πολιτικών αρχηγών ε, να μιλήσουν δημοσία υπέρ αυτών των ομάδων. Εάν βάλετε, δείτε στην ιστοσελίδα τι απαντήθηκε σε σχέση με αυτό το θέμα, βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιδράσεις μεταξύ των χωρών μελών και είναι ενδιαφέρουσες αυτές οι διαφορές. Ορισμένοι βλέπουν αυτή τη δυνατότητα και άλλοι όχι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της νομοθεσίας, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο που κατοχυρώνεται στο δίκαιο και στην εκπαίδευση η ίση μεταχείριση υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή για θέματα αυτά. Τώρα, όσον αφορά τους θήτες και τα περιστατικά βίας, ε, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες για τους δράστες και η εικόνα μάλλον δείχνει κάτι που γνωρίζουμε ήδη από άλλες έρευνες, ότι πολύ συχνά οι δράστες είναι νέοι άνδρες, καμιά φορά μεμονωμένοι ή και σε ομάδες και υπάρχει επίσης ένα θέμα ε, οικογενειακής ε, βίας, ε, πολύ ψηλά ποσοστά ανέφεραν περιστατικά βίας στο οικογενειακό περιβάλλον και έχουμε μια ανάλυση στη βασική μας έκθεση εν σχέση με το ποιοι είναι οι δράστες, ποιοι θεωρούν ότι είναι οι δράστες. Βέβαια πολύ συχνά δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι δράστες γιατί είναι περιστατικά που συμβαίνουν αργά τη νύχτα στο δρόμο. Αλλά κάτι ακόμα. Αυτές οι εμπειρίες των εγκλημάτων μίσου θα πρέπει να ειδωθούν κάτω από το πρίσμα των εκθέσεων της αστυνομίας. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα από τις ε, αρμόδιες αρχές όσον αφορά την ομοφοβική βία. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις για τους ΛΟΑΦ, ε, ούτως ώστε και οι αστυνομικές αρχές να μπορούν να είναι ανοιχτές στο να δεχθούν τέτοιου είδους καταγγελίες. Επίσης αναφέρθηκε από την κυρία Λούνατσεκ το θέμα γύρω από την ε, ταυτότητα φύλου, ε, το ζήτημα του ανδρισμού κλπ. Υπάρχουν ορισμένα ευρήματα τα οποία σχετίζονται πάρα πολύ με το φίλο. Δηλαδή όταν ρωτούμε πώς ε, αισθάνεστε, πώς εκφράζετε το φίλο σας, εδώ βλέπουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα ανάλογα με την ομάδα. Όσον αφορά η ανάγκη ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης, πράγματι είπαμε ότι υπάρχει μια ανάγκη οι χώρες μέλη να αντλήσουν δάγματα η μια από την άλλη, γιατί σε ορισμένες χώρες υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά το, ομόφοβο, το bullying λόγω ομοφοβίας, αλλά επίσης και στο επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης κλπ. και ε, των Ηνωμένων Εθνών υπάρχουν προπτικές συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και για την ε, συμμετοχή σας εδώ και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει μια παρακολούθηση των αποτελεσμάτων αυτής της έκθεσης του οργανισμού σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, ήρθε η κυρία Λίσβεκ, ε, οπότε προτείνω να προχωρήσουμε με μετά από μια πολύ σύντομη διακοπή. Uh, ε, μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Σημείο 19 της ημερήσιας διάταξης, η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στις 24 Απριλίου στη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ παρουσίασε η κυρία Γκρίσβεκ ε, το σχέδιο έκθεσης της 210 τροπολογίες ε, κατετέθησαν, ε, αν θυμάμαι καλά. Παρακαλώ όσοι αποχωρούν ε, από την αίθουσα, ας το κάνουν γρήγορα, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ένα λεπτάκι. have Όπως έλεγα, πάνω από 200 τροπολογίε. Έχουμε 210 συγκεκριμένα. Έγινε σύσκεψη σκιωδών ε, στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα και παρουσιάστηκαν και κάποιες συμβαστικές ε, τροπολογίες. Ε, στις 19 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η ψηφοφορία. Παρακαλούμε, κυρία Γκρίσβεκ, παρουσιάστε μας, αν θέλετε, τις συμβαστικές τροπολογίες και κάντε μας ένα απολογισμό των πεπραγμένων. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να συζητήσουμε για αυτήν την έκθεση για τους ασυνόδευτους ε, ανήλικους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να κάνω μία, ένα παρενθετικό σχόλιο προτού καταφτάσουμε και οι υπόλοιποι και αρχίσουμε να συζητούμε το ίδιο το θέμα για το χρονοδιάγραμμα και ακριβώς λόγω των πολυαριθμών τροπολογιών που έχουμε λάβει για το σχέδιο έκθεσης αποκτήσαμε έγινε δεκτή μάλλον η αίτηση παράτασης για την καταληκτική ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών. Δεν νομίζω να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Προτείναμε να συνεχιστεί η βάθος εργασία και να ψηφιστεί τελικά η έκθεση στις 19 και 20 του μήνα, αλλά ε, το απόγευμα στις 19 αντί για το πρωί, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά. Το είπατε λοιπόν ότι λάβαμε πάνω από 200 τροπολογίες για αυτό το κείμενο. Ε, φυσικά εγώ χαίρομαι διότι είναι ποικίλε οι απόψεις και μεγάλο το ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό. Αυτό καταδεικνύει ε, και τη σημασία αλλά και τον ευαίσθητο χαρακτήρα του ζητήματος στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σημερινή μέρα. Ως πλήστον εμπλουτίζεται η έκθεση με αυτές τις τροπολογίες, συμπληρώνονται κάποια στοιχεία. Στη σύσκεψη για τις συμβαστικές τροπολογίες, όπως μας είπατε, που έγινε ε, στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα, συζητήθηκαν επιμέρους ζητήματα και ε, με την ιδιότητα της εισηγήτριας ε, θα είναι μεγάλη μου χαρά ε, σε συνεργασία με τους αδέλφους να αποπειραθώ να καταλήξω σε κοινέ γραμμές κοινέ προσεγγίσεις και να προκύψει μια ενιαία θέση για αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που απέρριψα σχετικά γρήγορα. Είναι γλωσσικού χαρακτήρα αυτές οι τροπολογίες. Ε, συνάδελφοι, οι περισσότεροι καταθέσατε και τέτοιου είδους τροπολογίες, διότι υπήρξαν κάποια προβλήματα μετάφρασης. Ε, ε, μας εξέπληξαν εξάλλου στα αγγλικά, παραδείγματο χάρη, μιλάμε για overriding interest, αντί για best interest, που είναι η καθιερωμένη έκφραση. Αυτού του είδους οι τροπολογίες αυτή του είδους τροπολογίες επεξεργαστήκαμε και τις χτενήσαμε στη σύσκεψη των σκιωδών και αυτόματα δεχτήκαμε ε, όλοι ε, τις νέες τροπολογίες και ε, μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για ζητήματα τύπου αλλά και ουσίας γιατί οι γλωσσικές τροπολογίες δεν είναι θέματα τύπου είναι ζητήματα και πραγματικά ουσίας θα ήθελα, Πρόεδρε, να ασχοληθώ με τους βασικούς άξονες ε, της έκθεσης, ε, χρησιμοποιώντας ως γνώμονα ε, τις βασικές τροπολογίες ουσίας. Υπάρχει μια σειρά τροπολογιών που στόχο έχουν να προσθέσουν στοιχεία, να διευκρινίσουν τη διατύπωση, παραδείγματος χάρη τη νομική βάση του, του, που αναφέρεται στην έκθεση, τις διατάξεις που έχει ήδη αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό, δηλαδή το σύνολο των οδηγιών και κανονισμών, γενικές παρατηρήσεις της μόνιμης Επιτροπής για τα δικαιώματα των παιδιών, ε, ε, τον κανονισμό για την εμπορία των ανθρώπων που συζητήθηκε χτες στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όχι μόνο εμπλουτίζεται αλλά ολοκληρώνεται η έκθεση χάρη σε αυτές τις τροπολογίες. Είμαι επίσης πολύ θετικά διακείμενη σε σχέση με ε, τις τροπολογίες που προσδίδουν ένα νομικό βάθος ε, στην έκθεση για το θέμα της προστασίας των ανηλίκων, ε, τροπολογίες που αποσκοπούν στην καλύτερη οριοθέτηση ή την υπενθύμηση της αρχής που διέπει ε, ολόκληρη την παρουσίασή μου, δηλαδή το, ε, ε τον είπα στόχο μας, ε, τον ανώτατο στόχο μας, δηλαδή την προστασία των ανηλίκων. Αυτή ε, αυτή η καθοριστική αρχή επηρεάζει επίσης ε, μία σειρά διατάξεων για το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων ευρύτερα, αλλά και και εδώ πανεθετικά να πω ότι αυτό αναφέρεται σε διάφορες τροπολογίες ε, των συναδέλφων. Πρόκειται λοιπόν για τη διαπίστωση ότι τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία ή την ομολογία στον τομέα των συνόδευτων ανηλίκων και άρα ε, ο στόχος είναι να επιτύχουμε ορθότερη εφαρμογή και κυρίως ορθότερη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και υλοποίηση των ε, κείμενων διατάξεων προτείνεται διεξαγωγή πλήρους ε, αξιολόγησης συλλογικής και ατομικής, δηλαδή κατά περίπτωση, σε κάθε περίπτωση ανηλίκου. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Πέραν αυτού, ε, οι συνάδελφοι ασχολήθηκαν ναι, επισταμένα και με το άλλο εξίσου σημαντικό ζήτημα, κατάρτιση, επιμόρφωση των υπαλλήλων που καθημερινά ε, στη δουλειά τους έρχονται αντιμέτωποι με τους ασυνόδευτους ε, ανήλικους. Τώρα το άλλο ζήτημα είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών των ανηλίκων, οι όροι υποδοχής, πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνική ασφάλιση, στέγη, ε, ιατρικές υπηρεσίες και το καθεξής. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά και ε, ε, ενσωματώθηκαν στην έκθεση στις αποστολές που έγιναν κατά την προετοιμασία της έκθεσης σε διάφορα κράτη-μέλη, όχι σε όλα, αλλά σε διάφορα κράτη-μέλη μαζί με συναδέλφους, εφάνει πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε αυτές τις διαπιστώσεις, αλλά και στην Επιτροπή μας να καταλήξουμε σε μια συνενετική θέση. Είπαμε ότι έχουμε 210 τροπολογίες ε, με προτινόμενες διατυπώσεις για τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων. Προστασία των δεδομένων, ένα θέμα που αναφέρεται, ε, απαντάτε μάλλον στις παραγράφους όπου ε, πραγματευόμαστε το θέμα των στατιστικών στοιχείων, της ανάγκης συλλογής στατιστικών στοιχείων είναι αδύνατον να συγχέουμε τις ανώνυμες ε, ε, στατιστικές έρευνες με τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων. Ε, και είναι ένα θέμα ιδιαίτερα προσφυλές για την Επιτροπή μας. Όλοι επιθυμούμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τώρα, η... ως προς τον ίδιο τον ασυνόδευτο ανήλικα υπάρχει μια σειρά στοιχείων για τα οποία καταλήξαμε σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες για την εμπορία ανθρώπων, ε, αναφέρθηκα σύντομα σε αυτό, συγκεκριμένη προστασία ε, που χρήζει ο ε, κάποιος ασυνόδευτος ε, ανήλικος όταν πέφτει θύμα εμπορίας ανθρώπων. Συζητήσαμε χτες αυτό το ζήτημα με την κυρία Μύριαν Βασιλιάδου και θα ενσωματώσουμε αυτά τα στοιχεία επίσης πολυάριθμες. Επίσης ήταν τροπολογίες για το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων και ευελπιστώ ότι η συμβαστική στην οποία θα καταλήξουμε θα προσδώσει ε, συνοχή στην ε, έκθεση και θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε στη συμφωνία. Κάποιες ε, τροπολογίες όμως περιορίζουν το, κατά τι, το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού και υποβαθμίζουν την προστασία των ανηλίκων. Πάλι εδώ πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, παραδείγματο χάρη να καταστεί αδύνατη η κράτηση των ε, ανηλίκων. Νομίζω ότι είναι ένα, ε, μια κόκκινη γραμμή για την Επιτροπή μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια υποχώρηση ε, και να δεχτούμε διατάξεις που καθιστούν δυνατή την κράτηση των ανηλίκων. Για να μην πολυλογώ, θα ήθελα να υπενθυμίσω τους τρεις βασικούς άξονες που οπωσδήποτε θέλω να παραμείνουν μέσα στην έκθεσή μου και ε, ε, που συνιστούν και τον πυρήνα της πρότασης της έκθεσης πρωτοβουλίας που εξ ορισμού μας επιτρέπει όχι ε, να πούμε άνετα και να εκφράσουμε τα σώψυχά μας αλλά εν πάση περιπτώσει να τοποθετηθούμε με σαφήνεια και να πούμε αυτό που έχουμε να πούμε. Αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε και για συμβαστικέ τροπολογίε. Ένα, ε, στη διάθεση των κρατών μελών θα πρέπει να έχουμε ένα handbook, ένα εγχειρίδιο. Με τη Σεσίλια Μάλμστρομ το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και εκείνη μάλλον υπέρ. Ένα εγχειρίδιο λοιπόν όπου θα έχουμε τη συλλογή των νομικών βάσεων που είναι διάχυτε προ το παρόν ε, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που οι διατάξεις έχουν καταστεί δυσανάγνωστες πλέον. Ε, κατά τα λοιπά δεν υπάρχει κάποιο ρίξη και στοιχείο μέσα στο εγχειρίδιο, δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Κάνουμε μια απογραφή της κείμενης νομοθεσίας με αποδέκτες, με χρήστες αν θέλετε, τα κράτη-μέλη, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια ε, ως προς την νομοθεσία και να προσεγγίζουμε ορθότερα τη το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκτων. Δεύτερον, ε, η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ο στόχος μας είναι ε, να γίνονται σεβαστά τα ε, θεμελιώδη δικαιώματά τους σε όλα τα κράτη-μέλη. Πώς να το επιτύχουμε αυτό με τρόπο σαφή και εναρμονισμένο. Ε, λοιπόν, προτείνουμε να γίνει αυτό μέσω κατευθυντηρίων γραμμών, οι οποίες θα εδράζονται επί των βελτίστων πρακτικών των κρατών μελών και θα προτείνονται κοινά πρότυπα για κάποια ε, ζητήματα. Πέραν του εγχειριδίου λοιπόν και των νομικών βάσεων που υπάρχουν, θέλουμε να έχουμε ένα πρακτικό σημαντικό, εύχριστο, συνεκτικό εργαλείο στη διάθεση των κρατών μελών που είναι βασική εταίρη στη διαδικασία με στόχο να εφαρμοστούν τα ενιαία, τα κοινά ε, πρότυπα. Τρίτον, όπως σας είπα και προηγουμένως, αλλά ε, θα το ημεθυμίσω για να το εμπεδώσουν όλοι, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο ανήλικος είναι πάνω από όλα ή ένα παιδί ένας έφηβος και Άρα ανήκει σε ευπαθή, σε ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα και αυτή είναι η πρώτη βασική ιδέα. Και δεύτερη ιδέα, με διαρθρωμένο τρόπο θα πρέπει ε, σε σχέση με αυτά τα δύο εργαλεία να έχουμε πάντοτε κατά νου ε, την ίστατη ανησυχία, το ευζήν ε, του ανηλίκου είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε ε, μια τετράγωνη λογική και να ορίσουμε ε, τα συμφέροντα του παιδιού. Εγώ πραγματικά προβληματίστηκα πολύ στην αρχή και με ότι δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος ορισμός νομικός πώς όμως είναι δυσχερές να φανταστούμε στον ευρωπαϊκό χώρο ε, όλα τα παιδιά να εντάσσονται σε μια αυστηρή κατηγορία γιατί όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά και επίσης σε επίπεδο νομολογίας και νομοθεσίας ο ορισμός δεν υπάρχει, ε, ας το πω έτσι, στην νομοθεσία, υπάρχει μόνο στην νομολογία. Δεν θα ε, αρχίσω να εξετάζω μία-μία τις 210 τροπολογίες για θα τελειώσουμε αύριο, αλλά ήθελα μόνο να επιστήσω την προσοχή σας ε, στο ότι είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους για την έκθεση και ότι να τονίσω ότι ελπίζουμε πως ταχύτατα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες και μεταγενέσεις έστερα σε μια συνενετική θέση. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Ελπίζω, ε, χαίρομαι γιατί τώρα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Την τελευταία φορά δεν είχαμε καθόλου χρόνο. Ήθελα να ρωτήσω, να ζητήσω μάλλον από τους σκιώδεις εισηγητές να κάνουν σχόλια και μετά την ε, Κομισιόν, γιατί δεν είχε χρόνο η Κομισιόν την τελευταία φορά να κάνει σχόλια. Επομένως, η κυρία Κοράτσα Πιέρα. Ευχαριστώ. Ε, Κίνγκα, ευχαριστώ Ναταλή, να επαναλάβω για άλλη μια φορά τι, πόσο ευχάριστα ήταν να ε, δουλεύουμε μαζί και στην τελευταία φορά καταφέραμε στο Στρασβούργο να πετύχουμε πολλά πράγματα. Ε, δεν επαναλαμβάνουμε τα πράγματα, προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι. στην, στον πυρήνα των ανησυχιών μας έχουμε την, το παιδί και το πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε καλύτερα. Ε, η Κομισιόν θα δημιουργήσει αυτό το εγχειρίδιο για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το κατακαιρματισμό των νομικών κειμένων ε, και θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να συγκεντρώσουν όλες τις νομικές διατάξεις. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο είναι, και το αυτό το βάζω και στις τροπολογίες, θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν με ένα συνεκτικό τρόπο όλα τα ε, νομικά όργανα τα οποία υπάρχουν έτσι ώστε να έχουμε έναν πιο συνεκτικό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τους, τα, τους ασυνόδευτους ανήλικους και να ανεβάσουμε τα στάνταρτς για όλους. Ε, καλωσορίζω την ιδέα να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, δηλαδή να έχουμε ό,τι τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εκτίμηση της ηλικία, ε, ε, την ε, μεταβατική περίοδο, το παιδί όταν το παιδί γίνει 18, όταν γίνει ενήλικος, να εντοπίσει την οικογένειά του, το κηδεμόνας, ο δι, δι, διερμηνέας, ο νομικός εκπρόσωπος, για να ανεβάσουμε το επίπεδο, νομίζω ότι μπορούμε να δεχθούμε πολλά από τα άλλα κράτη-μέλη. Επίσης πρόσβαση στην, στις φροντίδες υγείας, στην εκπαίδευση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για έναν ασυνόδευτο ανήλικο. Επίσης ε, ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, ε, όταν συντάξαμε τις τροπολογίες. Να πω επίσης ότι πάρα πολλά νέα κορίτσια έρχονται στις χώρες μας ε, με τα παιδιά τους και αυτό είναι μια πρόκληση. Θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά αυτά με έναν ανθρώπινο τρόπο και διασφαλίζοντας ε, τα δικαιώματά τους. Μια και θα ψηφίσουμε τώρα τον Ιούνιο όλο το πακέτο για το άσυλο, όπου έχουμε συμπεριλάβει πολλά στοιχεία για την προστασία των ασυνόδευτων ε, ε, ανηλίκων να σας πω ότι δεν ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας ε, με, το, με την έκθεση αυτή ίσα ίσα ενισχύουμε το όλο οικοδόμημα, βοηθάμε τα κράτη-μέλη να διατυπώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την νομοθεσία. Επομένως, δεν θέλω σε αυτό το κείμενο να έχει κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία θα ψηφίσουμε στο πακέτο άσυλο και να σας να πω ότι ήταν ευχαρίστησή μου η συνεργασία με τους ε, ε, άλλους και Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την συνάδελφο την Ingrid ε, ήταν ε, η συνεργασία μας ιδιαίτερα επικοδομητική. Ε, αυτό ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, κυρίως όταν προσπαθείς να συμφιλιώσεις απόψεις που ενδεχόμενα να είναι αντιφατικές. Η Μπίλτη έκανε μια παρατήρηση, την οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Εφόσον το πακέτο άσυλο θα περάσει τον επόμενο μήνα, ε, αναφέρθηκε να πω ότι αποτελεί μία συμβιβαστική πρόταση ε, και βέβαια ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα συμβιβασμό θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, κυρίως όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Η συζήτηση αυτή όμως πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, διότι έχουμε μιλήσει ιδιαίτερα για τα δικαιώματα των, των ανθρώπων και μην ξεχνάμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα δικαιώματα αυτών των παιδιών που είναι η πιο ευάλωτη κατηγορία του πληθυσμού και πρόκειται για παιδιά που μπορεί να είναι και μετανάστες αλλά τέλος πάντων μιλάμε για άτομα τα οποία είναι κάτω των 18 δεν υπάρχουν ε, συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά το εύρος του προβλήματος. Ποιος είναι ο αριθμός των ε, παιδιών ή των νέων που μένουν ε, στις χώρες μας σαν ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε πιο αξιόπιστα στοιχεία. Αλλά ούτως ή άλλως τα στοιχεία αυτά πρέπει να συλλεχθούν για να προστατευτεί η κατάσταση των παιδιών και όχι για να δοθούν ε, στις δικαστικές αρχές. Επίσης, ε, θα πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα διακριτικοί, γιατί μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ε, για τις οικογένειες των παιδιών αυτών που έχουν μείνει στη χώρα τους. πρέπει να έχουμε τα στοιχεία για να ξέρουμε εάν ας πούμε η επιστροφή ε, στην χώρα του είναι μία λύση. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην, για να μην ε, αποτελεί κίνδυνο η επιστροφή αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει η οικογένειά του εκεί ή κάποιος τέλος πάντων να το υποδεχθεί και να μην λειτουργήσει εις βάρος του παιδιού η λύση αυτή. Επίσης, όσον αφορά το άσυλο, υπάρχουν ε, χώρες όπως η Γερμανία που μετέφερε την ε, οδηγία αυτή κατευθείαν στην ε, νομοθεσία ε, και εκεί στην οδηγία αυτή αναφέρεται και η ε, παράνομη διακίνηση των ατόμων. Επίσης, η πρόσβαση στο σχολείο, η πρόσβαση στις ιατροφαρμακευτικές, ε, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η στέγαση των παιδιών αυτών, των ασυνόδευτων. Δεν θα πρέπει να στεγάζονται τα παιδιά αυτά με ενήλικες. Θα πρέπει να τους ε, στεγάζουμε σε συγκεκριμένες ε, δομές. Ε, αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα πιστεύω ότι μαζί με, τον, ε, με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές ε, συμμεριζόμαστε έναν ενιαίο στόχο που είναι η προστασία των ασυνόδευτων ε, ανηλίκων. Ευχαριστώ. Η κυρία Φλότρο. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Ναταλή, διότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά που έκανε. Είχε έναν σαφή προσανατολισμό όσον αφορά την πρόκληση που παρουσίαζε η έκθεση αυτή, που ήταν να προστατεύσουμε τα, ε, τα, τα απομονωμένα παιδιά, ε, τα, τα, τα ανήλικα, τα οποία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν μετανάστες ε, έτσι ώστε να μην ε, συγκεντρώνουμε όλες τις ε, νομοθεσίες και να τις εφαρμόζουμε χωρίς να σκεφτόμαστε. Θα πρέπει η προσέγγιση όμως αυτή να γίνει σεβαστή, διότι μέσα από τις συμβαστικές προτάσεις συνειδητοποιούμε κάποια στιγμή ότι δίνουμε στην είσοδο, στην έξοδο και στην εργασία με τις τρίτες χώρες ένα, μια σημασία που δεν θέλαμε να δώσουμε στην αρχή. Επομένως, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τις δομές των κρατών μελών για να προστατεύσουν στην επικράτειά τους, τους, τα, τους ανήλικους ασυνόδευτους. Αυτό θα πρέπει να μην χαθεί κάπου στην πορεία. ούτως ή άλλως το θέμα είναι, είναι, το θέμα είναι τι θα δοθεί, τι ποιο θα είναι το νομικό βάρος, η νομική υπόσταση αυτού του κειμένου. Θα είναι κατευθυντήριες γραμμές, θα είναι σύσταση, θα είναι τι είναι. Α, τώρα έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Άρα ε, μπορούμε να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική ή αν δεν μας αρέσει η στρατηγική ποιος θα είναι ο τρόπος με τον οποίο προτίθενται τα κράτη-μέλη έτσι ώστε τα δικαιώματα, τα δικαιώματα των παιδιών για την υποδοχή, για την εκπαίδευση, για την υγεία, για την ε, ε, έρευνα της, για την οικογενειακή τους κατάσταση κτλ. Όλα αυτά να γίνουν σεβαστά. Τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη και πώς εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να ε, ελέγχουμε περιοδικά τι, τι γίνεται. Διότι αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Να έχουμε ένα κείμενο το οποίο να αναφέρεται όλο το, να αναφέρονται όλες οι διατάξεις ε, που θα επιτρέψουν σε κρατημέλη να κάνουν κάτι καλό. Αφενός, αφετέρου όμως εμείς θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική όπου να μπορούμε να ελέγχουμε τι προτίθεται να κάνουν τα κρατη και όταν μας λένε τι θα κάνουν τα κρατη να μπορούμε και εμείς να το ελέγχουμε ότι το έχουν κάνει. και θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς ε, να ευαισθητοποιούνται. Είτε πρόκειται για προστασία δικαιωμάτων γενικά, είτε προστασία των ε, δικαιωμάτων των παιδιών αφετέρου. Κατά δεύτερο λόγο, ο συσχετισμός μετανάστευση-ανάπτυξη νομίζω ότι κάτι, η κακή προσέγγιση είναι ή κακές προθέσεις είναι. Όταν αναπτύσσεται μία χώρα, ε, είναι δύσκολη, δεν, γίνεται, δεν υπάρχει μετανάστευση. Μετανάστευση από την χώρα. Και αυτό όμως δεν ισχύει, διότι πολλές φορές, έστω και αν υπάρχει ανάπτυξη, οι νέοι φεύγουν. Επομένως, ε, πολλά φορά, πολλές φορές κρύβουν, κρύβεται αυτή η αλήθεια. Και ένα το δεύτερον, που είναι κακή πρόθεση είναι να χρησιμοποιούμε τις πολιτικές ανάπτυξης ε, έτσι ώστε να ελέγχουμε τις χώρες προέλευσης, να εμποδίζουμε την ε, μετανάστευση. Γι' αυτό καλό θα είναι να καθαρίσουμε, αν θέλετε, αυτό το κείμενο, το κείμενο από, αυτές, από αυτό το συσχετισμό ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην ε, μετανάστευση. Επίσης, ε, οι, οι εκστρατείες πρόληψης της μετανάστευσης ε, ή κινδύνου της μετανάστευσης ε, είναι προσπάθειες να εμποδίσουμε τους ανθρώπους να φύγουν και αυτό είναι το αντίθετο από αυτό το οποίο θέλουμε εδώ στην Ευρώπη που λέμε στους νέους μας φύγετε, αποκτήστε νέες εμπειρίες, νέες ευκαιρίες. Επομένως αυτό το οποίο λέμε, δεν λέμε εδώ δεν μπορούμε να το λέμε σε τρίτες χώρες. Επομένω, και αυτή την αναφορά στην εκστρατεία πρόληψη θα ήθελα να ε, διαγράψουμε. Η, η αναφορά στην ε, επανεισδοχή Ακούσαμε τον κύριο Κρεπό για τα δικαιώματα των μεταναστών. Μίλησε για μεμονωμένους, απομονωμένους ε, ανήλικες. Ε, καμία κράτηση ανήλικου δεν μπορεί να είναι υπέρ του παιδιού είναι μία από τις συστάσεις που έκανε. Ταυτόχρονα αμφισβητούμε για τους ε, ανήλικους αλλά και για όλους ε, μέσα στα, στην επανεισδοχή να μην ε, σεβαστούμε τα δικαιώματά τους. Εγώ θα, θα έλεγα συγκεκριμένα οι ανήλικοι να συμπεριλαμβάνονται σε κάποιες συμφωνίες. Τώρα, όσον αφορά την επιστροφή, μήπως μπορούμε να είμαστε πιο απλοί. Μία επιστροφή Όντως, η επιστροφή μπορεί να είναι υπέρ του παιδιού, αλλά, αλλά ένα πρώτο τεστ θα ήταν πρέπει να συμφωνεί ο ανήλικος. Ίσως να μην αρκεί αυτό για να εξασφαλίσουμε ότι είναι υπέρ του, του παιδιού η επιστροφή, όμως αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει, αυτή η δικλίδα ασφαλείας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο. Είπα, είπα στην Αταλή ποιε είναι οι παρατηρήσει μου. Το μελετήσαμε, το μελέτησα πάρα πολύ και πιστεύω και την Αταλή θα τα λάβει υπόψη της όλα όσα είπα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήταν ουσιαστική η συζήτηση σε αυτό το θέμα. Ο κ. έχει το λόγο. Και εσείς επίσης. Σε λίγο. Δεν με πειράζει, λέει ο κύριο Τενταφυλλίδη. Τότε θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κίρκοπ. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο γιατί θα πρέπει να φύγω. Θα ήθελα καταρχήν να πω πόσο χρήσιμη ήταν η επίσκεψη της αντιπροσωπείας που είχαμε στη Σουηδία και θα ήθελα να μπουν στα πρακτικά, να, πει να αναφερθεί η γνωμοσύνη μου προς τις αρχές εκεί. Ε, ήταν πολύ χρήσιμη η εργασία μας εκεί. Θα ήθελα επίσης να στήσω συγγνώμη από την κυρία Γκρίσπεκ που δεν ήμουν σε θέση να πάω την προηγούμενη εβδομάδα στην συνάντηση, στη συνεδρίαση των σκιωδών γιατί είχα άλλε υποχρεώσεις, αλλά μου είπαν ήταν πολύ επικοδομητική και υπήρξαν πάρα πολλές συμβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να αναφερθώ στην 11 που αφορά την παράγραφο 14. Στη δική μου ε, στη δική μου τροπολογία στην παράγραφο 14, αναφέρω στις ε, ακτινογραφίες σαν ε, μη, δι, μη ε, βλαπτική μέθοδο ελέγχου. είναι σε σχέση με την ηλικία του παιδιού. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μνήα στην ε, ανάγκη να χρησιμοποιούνται ιατρικές μέθοδοι οι οποίες δεν είναι επιζήμιοι για την υγεία των παιδιών. Επίσης, η συμβαστική τροπολογία 6. Συμφωνώ επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων ε, για το σκοπό της προστασίας του, του παιδιού. Επίσης, η συμβαστική τροπολογία 10, ε, λέγοντας ότι η επίσημη διερμηνής δεν είναι πάντοτε αναγκαίο. Πιο σημαντικό είναι να υπάρχει κάποιος, ίσως και ένα μεγαλύτερο μέλος του προσωπικού που μπορεί να μιλήσει με το παιδί σε μια γλώσσα που να καταλαβαίνει το παιδί. Το να έχει κανείς ένα διερμηνία ενδεχομένω μια πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή ε, διαδικασία και ενδεχομένως μπορεί να καθυστερήσει την άντληση πληροφοριών για την πραγματική κατάσταση του παιδιού. Ε, θα ήθελα να πω ότι η ανθρωπιστική προσέγγιση που έχει πάρει η Σουηδία είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν θα πρέπει ε, ποτέ να επιτρέψουμε σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για αυτή τη, τα δεινά των παιδιών να υπεκφεύγουν τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν διεθνείς ε, διαβουλεύσεις ε, ούτως ώστε να ασχοληθούμε με μια πραγματικά ανήθικη ορισμένες φορές διαδικασία. Ορισμένες φορές υπάρχουν και εγκληματικέ προθέσεις και άλλες όχι. Οι ενήλικοι χρησιμοποιούν τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Ε, τα παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Τα παιδιά έχουν τα δικά τους δικαιώματα και χρήζουν προστασίας. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριο Τρενταφυλλίδη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και συμφωνώ με τον κύριο Κίρκοπ ε, εν σχέση με την ε, συνάντηση στην ε, Σουηδία. Ήταν πραγματικά η κατάλληλη στιγμή πριν από την συζήτηση εδώ αυτού του θέματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Γκρίσπεκ ε, που έχει μια πολύ γόνιμη προσέγγιση ε, και η συνάντηση που είχαμε στο Στρασβούργο ε, ήταν πραγματικά επικοδομητική. Τώρα όπως ακούσαμε υπάρχουν 210 τροπολογίες και αυτό είναι δεκτικό για, τις πολλές, για την πολυμορφία των απόψεων που έχουν διάφορες πολιτικές ομάδες και νομίζω ότι ενώ όλοι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ε, τελικά ε, είναι δύσκολο να βρεθεί μια κοινή λύση. Εγώ αναμένω με ενδιαφέρον τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές και ελπίζω τελικά να κατορθώσουν οι σκιώδεις να συγκεράσουν τις ε, διαφορές για να αποστείλουμε ένα χειρό μήνυμα προς την Επιτροπή και τις χώρες μέλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μπρόγκ έχει το λόγο. Ναι, έχω πολλές επιφυλάξεις σε σχέση με την ε, ιδέα ότι παιδιά 17 ετών έχουν τις γνώσεις και τη δυνατότητα να έρθουν στην Ευρώπη από άλλες υπήρους. Η ιδέα ότι οι νέοι άνθρωποι ε, οι άλλες ομάδες ανθρώπων το έκαναν στο παρελθόν δεν στέκει. Ε, εάν ε, ανήλικοι είναι πράγματι ασυνόδευτοι ε, όταν έρχονται στην προσοχή, υποπίπτουν στην προσοχή των αρχών, είτε υπήρξαν αντικείμενα διακίνηση από κάποιους εγκληματίες, οι οποίοι ασφαλώς θα πρέπει να διηθούν στη δικαιοσύνη ή συνοδεύονται από τις οικογένειές τους ή υπάρχουν οικογένειές τους κάπου που ήθελαν να τους στείλουν. Ε, και βεβαίως αυτό που καθορίζει την ε, απόφαση η οποία θα πάρθει. Ε, γιατί βεβαίως ένα παιδί στην Ευρώπη θα έχει καλύτερη εκπαίδευση και καλύτερη υγεία. Το ενδιαφέρον ως παιδιού να διαμείνει στη χώρα προέλευσής του, στη διευρυμένη οικογένεια, να, μιλήσει εκεί, να μιλάει τη γλώσσα του κλπ. Ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο συχνά παραμαλείται. Εδώ υπάρχει μία ατζέντα για περιόριστη μετανάστευση. Το μοντέλο των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι το τελευταίο κομμάτι αυτής της ε, πολιτικής. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Σμίτ, από την Κομισιό, να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Γκρίσμπεκ, για όλα αυτά που κάνατε, για το τόσο σημαντικό ζήτημα. Είναι εξαιρετικά επίκαιρο εξάλλου, διότι, όπως γνωρίζετε, παρουσιάσαμε το σχέδιο δράσης 2010 για τους ασυνόδευτους ανήλικους και πέρυσι είχαμε την έκθεση για την εφαρμογή της πρώτης διετίας ε, του σχεδίου δράσης εντοπίστηκαν κάποιες ελλείψεις οι οποίες καταγράφονται στην έκθεση και στις ε, άνω των 200 τροπολογίες ε, που έχουν κατατεθεί. Είναι, όπως πολλοί είπαν, εξαιρετικά λεπτό το ζήτημα αλλά και σημαντικό. Επίσης είναι εγκάρσιο διότι επισέρχεται σε διάφορες πολιτικές όλες τις διαστάσεις της μετανάστευσης, άσυλο, ενσωμάτωση η πιθανή επιστροφή. Ε, επίσης σχετίζεται με την εμπορία των ανθρώπων, συνεργασία με τρίτες χώρες. Ε, υπάρχει και το αναπτυξιακό κομμάτι, διότι συχνά οι νέοι που επιζητούν ένα καλύτερο τρόπο ζωής θα έπρεπε ε, ε, ιδανικά να ενισχύσουν την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε βεβαίως ε, ο βασικός νόμος είναι ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού, αν είναι η επιστροφή του στη χώρα προέλευσης ή η ενσωμάτωση στη χώρα υποδοχής. Ε, χρειάζεται συντονισμό ανάμεσα σε όλου αυτού του επιμέρου τομεί τη πολιτική και θα ήθελα να τονίσω ότι η εφαρμογή τη νομοθεσία ε, έχει μεγάλο ειδικό βάρο. Ε, θα έχουμε σύντομα το νέο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ΣΥΛΟΥ και σας διαβεβαιώ ότι θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς εξελίξης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα παρακολουθήσουμε όλες ιδιαίτερως τι διαστάσει αυτού του ζητήματο που σχετίζονται με του ασυνόδευτού ανηλίκου. Ε, πέρα από την εφαρμογή μιλάμε και για την ε, έμπρακτη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, διότι... Αυτό είναι ένα άλλο μήνυμα που θα πρέπει να περάσουμε ε, στην αυτό αρμοδιότητα των κρατών μελών και πέρα από την προστασία των παιδιών θα πρέπει να υπομισθούν την ευθύνη του και τα κράτη-μέλη και να εκτελέσουν τα συμπεφωνημένα. Σε σχέση με αυτές τις οδηγίες που αναφερθήκατε, θα ήθελα εγώ να σταθώ στην οδηγία για την επιστροφή. Εκεί σε διάφορα σημεία τονίζεται η σημασία της προστασίας ε, του παιδιού και του ανηλίκου που είναι ασυνόδευτος. Ε, ε, παρουσιάσαμε στο τέλος του 2013 ανακοίνωση για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή και πέραν αυτού θέλουμε να εξετάσουμε και τα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με τους ασυνόδευτους ανηλίκους, αν να εξετάσουμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα προστασίας και κυρίως να αντιμετωπίσουμε αυτό το ακαθόδε ζήτημα της κράτησης ε, των ανηλίκων ε, που ε, προς το παρόν δεν καλύπτεται στην οδηγία για την εμπορία των ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων. Υπάρχει σχετική οδηγία και την αναφέρατε κι εσείς. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και το παρακολουθούμε επίσης. Αυτή τη στιγμή γίνεται και μελέτη για μια άλλη οδηγία για την άδεια διαμονής για τα θύματα εμπορίας. Ε, εκεί θα εξετάσουμε πιο συγκεκριμένα την κατάσταση ε, που επικρατεί για τα παιδιά. Όλες αυτές οι συνιστώσεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ε, διαφάνεια. Χρειαζόμαστε ένα κείμενο, ένα εγχειρίδιο όπου θα ομαδοποιούμε τους κανόνες όταν έρχονται κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή όλοι αυτοί οι επιμέρους κανόνες των οδηγιών, των κανονισμών και ούτω καθεξής όταν καταφθάνουν και κατά την υποδοχή τους και σε μεταγενέστερη φάση κατά την ενσωμάτωσή τους ε, θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι κανόνες, ε, πώς ε, προστατεύουμε τα παιδιά και το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια αλλά και να επιτύχουμε μια ορθότερη εφαρμογή μέσω ενός τέτοιου εγχειριδίου. Ας περάσω σε κάποια άλλα ζητήματα που αναφέρθηκαν στην πιθανή εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών. Η Άσο ε, ε, έχει εργαστεί εντατικά ε, για αυτό το ζήτημα και πρέπει να ξέρετε ότι αναμένεται να εκδοθεί εγχειρίδιο από την Άσο για αυτό το ζήτημα τους επόμενους μήνες για την επανένωση των οικογενειών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την ζωή και εμάς. Είναι πολύ δύσκολο. Η κυδαιμονία είναι ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί πολλά κράτη-μέλη. Θα έπρεπε να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές σε αυτό το τομέα ε, καθώς και μια προϊόντα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για αυτό το ζήτημα. Α, τα δεδομένα. Πολύ σημαντικό. Ε, δεν έχουμε πάντα διαθέσιμα τα απαιτούμενα δεδο, στατιστικά στοιχεία. Τον Ιούλιο, σε συνέχεια του σχεδίου δράση, ε, η Eurostat θα μας προσκομίσει τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία, απαιτούμενα για την πλήρη κατανόηση όλων των διαστάσεων του ζητήματος. Όλα αυτά θα πρέπει να συμβούν σε πλήρη σεβασμό των συμφερόντων των παιδιών βάσει και του σχεδίου δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε, βασιζόμαστε επίσης ε, σε μεγάλο βαθμό στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών και σε αυτό που έχει κάνει, είπατε, η αρμοστία του ΟΗΕ για τον προσδιορισμό ακριβώς των αναγκών των παιδιών και των συνοδευτών ανηλίκων. Δεν πρέπει να έχουμε πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς ανά θεσμικό όργανο ή ανά εθνική αρχή και το έρισμα όλων των δράσεων είναι το ε, καλύτερο συμφέρον του παιδιού. Ε, είναι πολύ επίκαιρο το ζήτημα λοιπόν. Το σχεδίο δράσης θα ολοκληρωθεί το 2014. Θα αντλήσουμε διδάγματα από την εφαρμογή του πρώτου σχεδίου δράσης. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, θα εξετάσουμε τι, ε, που επιδέχεται βελτιώσεις, για το άσυλο και τη μετανάστευση ενδέχεται να λάβουμε και χρηματοδοτική Υπάρχει φυσικά το Ταμείο για την ε, ε, ένταξη των ε, μεταναστών. Θα δούμε στο μέλλον πώς θα διαμορφωθεί η χρηματοδότηση. Έχουμε και πιλωτική δράση που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την... τους ασυνόδητους ενηλίκους και συνεχίζεται η δουλειά για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαστε εδώ για να υποστηρίσουμε το έργο σας ως συνήθως. σε ευχαριστώ. Ναταλή Γκρισμπέκ για τα καταληκτικά σχόλια. Euh, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους αλλά και στην Κομισιό που έκανε τα σχόλια αυτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω συγκεκριμένα τους συναδέλφους διότι η δουλειά ήταν πάρα πολύ σημαντική, δεν ολοκληρώθηκε βέβαια αλλά πιστέψω, πιστεύω ότι πάνω σε αυτό το θέμα που είναι ένα θέμα όπου δεν είναι και προφανές ότι θα συμφωνήσουμε. Ε, οι θέσει ε, δηλαδή που ακούγονται μπορεί να είναι διαφορετικές ή τουλάχιστον δεν είναι κοινέ. Ε, δεσμεύομαι να συνεχίσω την προσπάθειά μου να καταλήξω σε κάτι, σε ένα κείμενο που να είναι ικανοποιητικό και που να εξυπηρετεί τον κοινό μας στόχο. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια αυτό το σημαντικό θέμα. Διότι είναι ένα θέμα σημαντικό και για τα κράτη-μέλη, αλλά και για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χωρίς να χρονοτριβώ να σας πω ότι κατέγραψα όλα τα σχόλια και εάν ξέχασα κάτι, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, θα επανέλθουμε ε, στη συνέχεια των εργασιών για την ε, ερώτηση της Άννας Μαρίας να πω ότι η, δίνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρουσία των κοριτσιών, των ασυνόδευτων κοριτσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπενθύμησε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο πάνω στο οποίο όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμοστούν όλα αυτά και από τα κράτη. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει και μια ισορροπία με το ευρωπαϊκό σχέδιο. Ε, ε, ευχαριστώ και τους άλλους συναδέλφους για τον όρο παιδί. Ε, θεωρήσαμε ότι καλύτερα είναι να πούμε παιδί και όχι ανήλικος. Περιμένουμε από την νομική υπηρεσία να μας πει αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο παιδί για τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία. Όλοι συμφωνούμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία τα οποία να είναι πιο αξιόπιστα και να μην χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους παρά μόνο για την προστασία των ανηλίκων. Στην Ελέν Φλότχο, την οποία ευχαριστώ για την τόσο ε, ζωντανή της ε, ε, και θρηλυκή ζωτικότητα και ενέργεια με την οποία απαντά, όντως υπάρχει αυτή η ισορροπία μετανάστης παιδί ε, νομίζω ότι υπάρχει αυτή η ισορροπία, δηλαδή θα, προσπαθούμε να το, θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα των ανηλίκων θα πρέπει να υπάρχει πάντα στους διαλόγους που η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει με, τους, με τις τρίτες χώρες. Και το θέμα της... Ε, ε, παρουσίας των ασυνόδευτων ανηλίκων ε, συμπεριλαμβάνεται και στις συζητήσεις ε, που έχει η Ένωση με τις τρίτες χώρες για τα θέματα ανάπτυξης. Και πιστεύω ότι αυτό το θέμα, να μην το πω πρόβλημα, θα πρέπει να συζητείτε με τις τρίτες χώρες, με τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Βέβαια το άρθρο 7 θα το βελτιώσουμε για τα θέματα επανεισδοχής. Οι συμφωνίες επανεισδοχής υπάρχουν, άρα θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχει μια πραγματική προστασία και οι εγγυήσει ε, σε σχέση με τα θέματα αυτά. Μετά, όσον αφορά ε, τα σχόλια που έκανε η Ελέν Φλότχα, για το handbook ε, και τις κατευθυντήριες γραμμές εγώ είμαι σαφής υπάρχει από τη μια πλευρά η απογραφή όπως είπαν και οι συναδέλφοι, οι συνάδελφοι και η εκπρόσωπος της Κομισιόν και μετά υπάρχουν οι κατευθυντήριες γραμμές ε, πάνω στις οποίες συμφωνούμε και τις οποίες πρέπει να εφαρμόσουμε. Εγώ δεν χρησιμοποίησα τον όρο στρατηγική γιατί πιστεύω ότι ο όρος στρατηγική όταν χρησιμοποιείται για κάποιες στρατηγικές στην Ευρώπη στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμογής αυτής της στρατηγικής ε, τα αποτελέσματα δεν ε, φαίνονται τουλάχιστον. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προτίμησα τον όρο κατευθυντήριες γραμμές. Από την άλλη πλευρά μου άρεσε πολύ αυτό το οποίο ελέγχθη με το task force, δεν είναι πολύ καλά τα αγγλικά μου αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω, για να ελέγξουμε αυτό το οποίο κάνουν τα κράτη-μέλη. Δηλαδή να υπάρχει μια, ένας απολογισμός και να ε, μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε το δικό μας εργαλείο για να ζητήσουμε τον έλεγχο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και ελπίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία. Για την επανεισδοχή είπαμε, για την ε, κυρία Κίρκοφ να πω ότι την ευχαριστώ που μας ευχαρίστησε για την αποστολή στην Σουηδία. Για τους διερμηνείς θα βρούμε μια συμφωνία. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ο νέος να μπορεί να καταλάβει και να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του ή μια γλώσσα του, η μια γλωσσα η οποία, την οποία κατανοεί στη Σουηδία. Είδαμε ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Το ουσιαστικό είναι ο νέος να καταλαβαίνει, το παιδί να καταλαβαίνει και να κάνει διάλογο. Τώρα για το καθορισμό της ηλικία είδαμε διάφορους τρόπους ε, υπολογισμού που είναι ε, κατά την άποψή μου κατακριτέοι, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να τους υιοθετήσουμε, αλλά τέλος πάντων ο καθορισμός της ηλικία θα πρέπει καταρχάς να γίνεται με μεθόδους που να είναι λογικές και να, είναι, ε, να στηρίζονται στην, στον σεβασμό ε, του, και στην αξιοπρέπεια του ενδιαφερομένου, δηλαδή του παιδιού και να, να λαμβάνουμε υπόψη μας το ευάλωτο χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας. Τον Κυριάκο τον ευχαριστώ για όλη τη δουλειά που έκανε, για τις σκέψεις του, για την ε, διπλωματική του προσπάθεια. Νομίζω ότι όλοι συμφωνήσαμε να υπενθυμίσουμε και να υπενθυμίσουμε την ε, ε, τη χρήση των στοιχείων ε, και την ε, πρόσβαση σε πληροφορίες. Άκουσα τον συνάδελφο Μπρόνς με προσοχή και ευχαριστώ επίσης και την Κομισιό για τις διευκρινήσεις που έκανε για την οδηγία για την επιστροφή, για την διαφάνεια και χαίρομαι γιατί Ε, βλέπω στην Κομισιό μία ε, φροντίδα και, μία, και ένα στήριγμα. Τώρα για το πακέτο άσυλο. Όλοι χαιρόμαστε που επιτέλους ε, θα προσγειωθεί, αλλά εάν δεν προχωράει τόσο πολύ όσο εγώ προτείνω για την κράτηση, παραδείγματος χάρη, αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοώ τι υπάρχει στο πακέτο για το άσυλο, αλλά στην έκθεση πρωτοβουλίας, ιδίας πρωτοβουλίας, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, ό,τι επιθυμούμε. Άρα δεν υπάρχει αντίθεση κατά την άποψή μου. Δεν επηρεάζεται το έργο της Επιτροπής από το περιεχόμενο του πακέτου για το άσυλο. Λοιπόν, θα επανέλθω, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, Ευχαριστώ όλους και τους κοιόδης εισηγητές ε, για την ε, συνέπειά τους, για το χιούμορ που έδειξαν, που μας επέτρεψε να προχωρήσουμε. Γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν είμαστε από την αρχή όλοι σύμφωνοι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ επίσης πολύ και για την ε, συζήτηση και όπως είπαμε η ψηφοφορία θα γίνει στις 19 Ιουνίου. Τώρα έχουμε άλλο ένα σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα το πρωί που είναι η εφαρμογή της οδηγίας του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Ε, συντάκτης γνωμοδότησης είναι ο Ραούλ Ρωμέβα Ιρουέδα και θα του ζητήσουμε να παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης είναι μια γνωμοδότηση για μια έκθεση διας ε, πρωτοβουλίας της ε, Επιτροπής ε, Απασχόλησης εν σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας. Υπάρχει μια κίνηση στην αίθουσα. Θα έχουμε κάποιο χρόνο για σχόλια και από τους σκιώδεις. Κύριε Ρωμέβα, παρακαλώ, έχετε το λόγο και θα ήθελα να ζητήσω και πάλι από αυτούς που εγκαταλείπουν την αίθουσα παρακαλώ να το κάνουν με ησυχία για να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο επαναλαμβάνεται στις τελευταίες συζητήσεις και εδώ και τέσσερα χρόνια επιμένουμε το θέμα αυτό της ε, άνησης μεταχείρισης και των διακρίσεων εκτός της απασχόλησης παραμένει ένα από τα θέματα τα οποία επιδέχονται βελτιώσει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και στο μέτρο αυτό ήταν ότι υποφεληθήκαμε επίση από την ευκαιρία που υπάρχει αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας στην Επιτροπή Απασχόλησης για να υπενθυμίσουμε ότι ε, θα πρέπει τουλάχιστον ε, τα τέσσερα σημεία τα οποία είναι για μας σημαντικά να συμπεριληφθούν. Ε, πρωτίστως, ε, στη δική μας γνωμοδότηση, αυτό το οποίο θέτουμε στην έκθεση πρωτοβουλίας είναι να επισημάνουμε με τρόπο ρητό την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κά κάποιος εκτός εργασίας ε, σήμερα δεν προστατεύεται εάν υφίσταται διακρίσεις για λόγους θρησκευτικών πεπιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Αυτά τα, αυτές τις τέσσερις πτυχές ε, παραμένουν εκτός του χώρου εργασίας και οι διακρίσεις αυτές είναι μόνιμο φαινόμενο, το έχουμε δει άλλωστε ε, κατά επανάληψη σε διάφορες εκθέσεις και θα έχουμε μελλοντικά και περισσότερες αποδείξεις ότι η κατάσταση αυτή, υπό την έννοια αυτή, είναι ανησυχητική υπάρχει ένα περιβάλλον προστασίας στο χώρο εργασίας, αλλά όχι εκτός αυτού στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Εκπαίδευση, πρόσβαση στις υπηρεσίες, κοινωνική προστασία κλπ. Θέλαμε λοιπόν να καταγγείλουμε αυτή την έλλειψη. Και είναι σημαντικό στο μέτρο που αυτή η κατάσταση είναι καλά καλυμμένη σε ορισμένες χώρες μέλη, αλλά όχι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Αυτή είναι η πρώτη βασική ιδέα που θέτουμε στην γνωμοδότηση. Η δεύτερη είναι ε, επί της ουσίας ε, σχετίζεται με την ανάγκη να κατανοήσουμε ως βασική αρχή το αδιέρετο και το αναπαλωτρίωτο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ε, καθολικότητα και το αδιέρετο, το αναπαλωτρίωτο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην ε, σχέση, στη συνάφεια μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό σε Ευρωπαϊκή Ένωση να, να διαδώσουμε προς τα έξω αυτή την βασική ιδέα ότι τα δικαιώματα δεν, είναι, δεν πρέπει να διαιρεθούν ε, να διασπαστούν, αποτελούν ενιαίο σύνολο το οποίο θα πρέπει να υπερασπιστούμε ως σύνολο και υπό, το την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες ε, περιοχές ε, ορφανές εγγύησεων και προστασίας, αυτό είναι ένα έλλειμμα το οποίο θα πρέπει να διορθώσουμε. Και αυτό είναι ένα από τα αιτήματα που θέτουμε στην πρόταση γνωμοδότησης. Επίσης, υπάρχει μια ρητή ανάγκη να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να απαγορεύει ορισμένα κενά από αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε διάφορες χώρες ακριβώς λόγω έλλειψης αυτού του νομικού πλαισίου. Η τρίτη ιδέα που θέλουμε να θέσουμε είναι εξή. Θα υψώσουμε λίγο τον τόνο. Ε, δεν θα σας ε, διηγηθώ τις απογοητεύσεις που έχω αισθανθεί εδώ και τέσσερα χρόνια σε σχέση με το θέμα αυτό. Ε, το Συμβούλιο, δηλαδή οι κυβερνήσεις, ολιγορούν περιμένουμε να ολοκληρώσουν τη δική τους εργασία σε σχέση με την οδηγία, αλλά δεν το κάνουν. Υπάρχει βέβαια κάποια κίνηση εντός του Συμβουλίου και ορισμένες προεδρίες, άλλες πιο δυναμικά, μερικές πιο δυναμικά από άλλες, ε, μπόρεσαν να εργαστούν και να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες στο επίπεδο ορισμένων χωρών, αλλά από την άλλη ακόμα υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία μπλοκάρει την κατάσταση και εμποδίσει το Συμβούλιο να παρουσιάσει την πρόταση στο Κοινοβούλιο του, ώστε να μπορέσουμε εμεί να κάνουμε τη δική μα εργασία σε συνάρτηση ακριβώ με το κείμενο το οποίο θα μα παρουσιάσουν. Και εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη και προφανή δυσκολία με έλλειψη πολιτική βούληση. Είναι μια ξεκάθαρη έλλειψη πολιτική βούληση. Και εγώ θα έλεγα ε, μάλιστα κατάχρηση αν θέλετε της αρχής της ομοφωνίας εντός του Συμβουλίου. Περί αυτού πρόκειται. Και υπό την έννοια αυτή ε, θα πρέπει να βάλουμε το Συμβούλιο ε, ρητά, να ζητήσουμε να είναι σε θέση να, απομπλοκάρει αυτή την, να ξεμπλοκάρει αυτή την κατάσταση. Ε, υπάρχουν σε χώρες όπου υπάρχουν σοβαρές ε, αντιστάσεις όπως είναι η Γερμανία. Η, Γερμανία η γερμανική κυβέρνηση είναι αυτή που μπλοκάρει το θέμα αλλά ελπίζουμε ενδεχομένω ότι με μια αλλαγή της ε, κυβέρνησης ε, να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, είναι σημαντικό και αυτή είναι η τέταρτη σκέψη να επενθυμίσουμε κάτι το οποίο για μένα είναι θεμελιώδες ιδιαίτερος στο πλαίσιο των προσεχών εκλογών του 2014. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 12 φορές ζήτησε από το Συμβούλιο να απεμπλέξει την κατάσταση σε, βάρια, ε, σε, σε, διάφορα, ε, σε διάφορες συγκυρίες, διαφορετικά μεταξύ τους πλαίσια έχουμε επιμείνει. Η βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ξεκάθαρη. Ε, είναι ξεκάθαρη λοιπόν η πρόθεση του οργάνου που εκπροσωπεί τους πολίτες και από άποψη ευρωπαϊκής αξιοπιστίας πρόκειται για ένα ουσιαστικό θέμα το οποίο θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής ε, των ευρωεκλογών γιατί συναρτάται ακριβώς με το δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο μας ανησυχεί εδώ. Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές ε, σκέψεις που συμπεριλήφθηκαν από τον ε, συγητή τον κύριο, επί της ουσίας τον κύριο Κώσα στο βασικό του κείμενο. Νομίζω ότι η ευσεβής πόθη είναι το καλύτερο εδώ σε αυτή την περίπτωση. Η Έντιθ Μπάουρ ζήτησε το λόγο. Ο κύριος Κόσα εξέταζε τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η νομοθεσία με βάση τις ε, αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το να κατηγορήσουμε, να ανακατηγορούμε την οδηγία ότι δεν αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα. Ίσως να είναι και δικαιολογημένο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ε, για να προχωρήσουμε, διότι ο στόχος της οδηγίας για την απασχόληση είναι περιορισμένος. αλλά δεν είναι τόσο όσο τον αναφέρει ο εισηγητής. τα σωματεία, τα συνδικάτα, ε, η επαγγελματική κατάρτιση. Είναι σοβαρά, είναι σημαντικά θέματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία συμπληρωματικά σε σχέση με αυτά τα οποία συμπεριέλαβε ο εισηγητής της προτάσεις. Το ένα είναι τα νομικά βοηθήματα, η Κομισιό πρότεινε να, ότι θα υπέβαλε, μας είχε πει μάλλον ότι θα, θα υπέβαλε ένα κείμενο για, την συλλογική, για, το, για συλλογικά νομικά βοηθήματα μέχρι το τέλος ε, της προηγούμενης ε, χρονιάς. Αυτό όμως ακόμα περιμένει πρόβλημα. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι φορείς ε, ε, ίσων ευκαιριών εργάζονται με διαφορετικά, ε, διαφορετικές εντολές και η νομολογία των δικαστηρίων είναι διαφορετική στα κράτη-μέλη, Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον ο οποίος έχει υποστεί διακριτική μεταχείριση να στραφεί προς τα δικαστήρια, γιατί οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές. Αλλού χρειάζεται να πληρώσει κάποια προκαταβολή. σε άλλες χώρες είναι ελεύθερη η προσφυγή στα δικαστήρια. Υπάρχουν τέτοιου είδους διαφορές τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Τώρα, όταν η οδηγία αυτή υιοθετήθηκε το 2000, το άρθρο για την διακριτική μεταχείριση στη συνθήκη αναφέρονταν σε 8 κριτήρια. Η οδηγία αναφέρεται σε 5. Η χάρτα τώρα θεμελιωδών δικαιωμάτων αναφέρεται σε 16 κριτήρια. Τι θα γίνει με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε. Θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση, διότι ο κανόνας για την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης είναι ένας κανόνας, ο οποίος, μια διάταξη, η οποία θα στηρίζεται στο χάρτη και ε, εκεί αναφέρονται 16 κριτήρια. Άρα υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αλλαγές. Εγώ θα καταβάλω κάθε προσπάθεια η Σοφή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και στον εισηγητή για, την, για το κείμενο. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες για να ενισχύσω τα σημεία τα οποία έκανε, γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί του και συμφωνώ και με αυτά που είπε η κυρία Μπάουερ επίσης κατά πολύ, διότι έθιξε μερικά πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Αλλά όμως όταν μιλάμε για διάκριση στον χώρο εργασίας πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Η έκθεση η οποία μας, μας ε, ε, παρουσιάστηκα σήμερα για την ε, διακριτική μεταχείριση των λεσβιών, ομοφιλοφίλων και λοιπόν στο χώρο εργασίας δείχνει ποια είναι η πραγματικότητα. Δεύτερον, θα πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλά ή κάποια κρατημέλη τουλάχιστον όχι απλώς και μόνο μπλοκάρουν την ε, υιοθέτηση της οδηγίας, ίσα ίσα ε, νομοθετούν ε, με βάση κριτήρια διάκρισης. Δεν χρειάζεται να πούμε ποια είναι τα κράτη-μέλη αυτά. Είναι ένα κράτος το οποίο θα, γίνει, θα αναλάβει την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σονούπο και υιοθετεί νομοθεσία κατά των ομοφιλοφίλων προς, ε, υιοθέτησε πρόσφατα. Τώρα, επίσης στη Γερμανία, ε, όπου έχει θεσμοθετηθεί, είναι νόμος η διακριτική μεταχείριση με βάση την θρησκευτική, θρησκευτικές πεπιθήσεις. Η, η Εκκλησία είναι ο δεύτερος εργοδότης, ο μεγαλύτερος εργοδότης στη Γερμανία και έχουν τους δικούς τους ε, εργατικούς νόμους. Επίσης, έχει, τώρα έχει υποβληθεί ε, μία νομοθετική πρόταση για να αλλάξει αυτό. Αλλά ε, είναι θεσμοθετημένη η μεταχείριση, η διακριτική μεταχείριση για άτομα τα οποία δεν ε, δέχονται το ήθος ε, της εταιρεία ε, γιατί είναι ομοφιλόφιλοι, γιατί δεν ξέρω και εγώ τι, για λόγους τέλος πάντων που δεν έχουν να κάνουν με την δουλειά αλλά με την προσωπική του ζωή και αυτό είναι σαφέστατη παραβίαση των ελευθεριών των ατόμων. Και ήδη τώρα γίνεται μια κίνηση από πλευρά των συνδικάτων, ελπίζω ότι θα προχωρήσει. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ε, ότι αυτές είναι οι τροπολογίες που θέλω να υποβάλω ε, σε αυτούς το τομείς. Ε, θα πρέπει να σταματήσουμε να εκφράζουμε μόνο ευσεβείς πόθους και θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μπορεί το ένα κράτος μέλος να κρύβει το άλλο. Όλοι μιλάμε για τη μη διακριτική μεταχείριση και για τις ευρωπαϊκές αξίες και ιδιώδη. Είναι όμως όλα λόγια. Μήπως θα μπορούσαμε να το πούμε καθαρά όλους, σε όλους και να πούμε στους πολίτες ότι εμείς θέλουμε να έχουμε ε, ίσα δικαιώματα, αλλά τα κράτη-μέλη δεν το θέλουν, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ. Σήμερα ε, όλο το πρωί ασχοληθήκαμε αυτές τις συγκρούσεις λεκτικά, λεκτικά μηνύματα από τη μια και πραγματικότητα από την άλλη. και όσοι ήταν εδώ όλο το πρωί τα πήραν τα μηνύματα αυτά. Δεν βλέπω να θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Επομένως, θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ρωμέβα να σχολιάσει. Ευχαριστώ πολύ. Α, περιμένω με ανυπομονησία τις τροπολογίες. Πολλά από όσα θα περιλαμβάνονται ε, θα τα ε, ενδεχομένως ε, θα τα έχω ήδη συμπεριλάβει θα, ή μάλλον θα χαρώ πάρα πολύ να τα συμπεριλάβω. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Το ένα αυτό που είπε η κυρία Μπάουρ, το νομικό επίπεδο. Εδώ έχουμε κάποιες εμπειρίες και μπορούμε να αποδείξουμε πόσο σημαντικό είναι Ορισμένοι θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι παχθές. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι και να μην υπάρξουν εξαιρέσεις από το φάσμα εφαρμογή. Όσον αφορά τα σχόλια της Σόφη, είναι σημαντικό να μείνουμε στο εξή. Ε, ε, γνωρίζω ότι το αρχικό κείμενο είχε να κάνει με τις διακρίσεις εντός του χώρου εργασίας. Αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συνεκτική πολιτική κατά των διακρίσεων εάν δεν απαλληφθούν οι διακρίσεις όχι μόνο εντός του χώρου εργασίας αλλά και εκτός σε όλους τους τομείς. Επιθυμούμε λοιπόν να διευρύνουμε αυτό το πεδίο συμπεριλαμβάνοντας και άλλες σφαίρες της ζωής μας. Ε, πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες, κοινωνική προστασία κλπ. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρξει αυτή η διάσταση. Και ψώνοντας τη φωνή μας, είναι αναγκαίο, συμφωνούμε απολύτως. Ο κίνδυνος αναθερθούμε ότι είμαστε βόντες εν τη ερήμου. Και ενδεχομένως ε, θα υπάρξουν αρνητικές ανδράσεις αν ε, δεν υπάρξουν απτά αποτελέσματα. Γιατί αν κάποιος μας ρωτήσει τι θα πάρετε συγκεκριμένα, θα κερδίσετε συγκεκριμένα από όλο αυτό. Ε, σε τι χρησιμεύετε τελικά ως βουλευτές αν δεν ε, καταλήγετε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτή τη στιγμή ε, έχουμε τις τροπολογίες, θα ξεκινήσουμε με την επεξεργασία. Η ημερομηνία για την κατάσταση τροπολογιών είναι 10 Ιουνίου, Δευτέρα. Ολοκληρώνεται εδώ η πρωινή μας συνεδρία. Σε ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχατε και θα βρεθούμε στις 3 ε, το απόγευμα.